Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Να ξεκινήσουμε, να πάμε στο σημείο της ημερησίας διάταξης, στο σημείο 8, ε, ο προϋπολογισμός του 2014 και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο Γιώργο Σταυρακάκη να μας παρουσιάσει την ε, γνωμοδότησή του. ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την εισηγήτρια για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014, την Άννα Αναγκέσεν, στην Επιτροπή μας. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Γενικού Εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των μελών των επιμέρους των ειδικευμένων επιτροπών κρίνεται ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει στο Γενικό Εισηγητή να αποκτήσει μια σφαιρική άποψη των ζητημάτων που απασχολούν την εκάστοτε Επιτροπή. Και φυσικά δεν πρόκειται να αποτελέσει έκπληξη στην κυρία Γένσεν ότι το κύριο ζήτημα που απασχολεί την Επιτροπή μα είναι το επίπεδο πληρωμών, level of payments, στην πολιτική συνοχή. Σε αυτό το σημείο θα με επιτρέψετε να μην σα περιγράψω παράγραφο προ παράγραφο το τι περιέχει το σχέδιο γνωμοδότηση, εξάλλου το έχετε όλοι μπροστά σα. Ωστόσο, θα ήθελα να εστιάσω στο διαδικαστικό τη υπόθεση. Όλοι σα γνωρίζετε πολύ καλά πώ έχει η κατάσταση η Επιτροπή έχει καθυστερήσει την έκδοση του σχεδίου προπολογισμού για το 2014, το οποίο πλέον αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του Μαΐου. Επίσης, ελλείψη συμφωνίας για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 δεν γνωρίζουμε τα ανώτατα όρια των δαπανών για το 2014. Και συμφωνώ ότι χωρίς να έχει καθαριστεί πρώτα το ζήτημα με τα συσσωρευμένα αιτήματα πληρωμών, accumulated payment ε, claims, από τα προηγούμενα έτη, οι διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό του 2014 θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι όπως δήλωσε ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 13ης Μαρτίου για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να αποφύγουμε περαιτέρω μεταφορές των πληρωμών από το 2013 στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως καταλαβαίνετε, υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, η εκπόνηση του σχεδίου γνωμοδότηση από μόνη τη ήταν μια πρόκληση. Γι' αυτό το λόγο το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης που έχετε στα χέρια σα είναι όσο το δυνατόν πιο γενικό γίνεται. Συνεψίζοντα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στόχο μα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση ενό ικανοποιητικού επίπεδου χρηματοδότηση, το οποίο θα εξασφαλίζει του στόχου τη πολιτική συνεχή και την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων τη, ιδιαίτερα εν ώψη τη νέα προγραμματική περίοδου. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για να υποβάλλετε τις προτάσεις στη Γραμματεία σχετικά με τα πιλωτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που θα προτείνει η Επιτροπή μας είναι στις 8 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. We have... Ευχαριστώ. Ο κ. Γιάννης είναι ο για τον προϋπολογισμό τη Επιτροπή Προπολογισμών. Ο αρμόδιο δηλαδή τη Επιτροπή Προπολογισμών και είναι εδώ. Σα ευχαριστώ που ήρθατε, κυρία Γένσεν. Ε, μπορεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σταυρακάκη για την παρέμβασή του. Όντως, ειδικά για την περιφερειακή πολιτική, η κατάσταση είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Θα θυμάστε ότι το Μάρτιο ψηφίσαμε ε, κατευθυντήριε γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014. Οι κατευθυντήριε γραμμές διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες. καταρχά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν έχουμε δηλαδή τη νομική βάση για τον προπολογισμό ή το πλαισιο προπολογισμου προϋπολογισμού 14-20. Υπάρχει γενικό πρόβλημα, αλλά ακόμα περισσότερο στις περιφερειακές πολιτικές. Δεύτερον, το θέμα των πληρωμών. Το πρόβλημα είναι όλο ένα και πιο έντονο, γιατί το Συμβούλιο δεν θέλει να πληρώσει λογαριασμού. Δεν θέλει να καταβάλει τα λεφτά που χρειάζονται για τις απαιτήσει που υπάρχουν. Και πουθενά αυτό το πρόβλημα δεν είναι πιο οξύ από ό,τι στην περιφερειακή πολιτική. Τέλος. Αναφέραμε τις πολιτικές προτεραιότητες για το 2014, όπου το, το Κοινοβούλιο συμφώνησε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενεργεία των νέων. Έχουμε την πρωτοβουλία για τους νέους, την επερχόμενη, και βεβαίως τη στρατηγική του 2020 που είναι το γενικό πλαίσιο. Όμως η περιφερειακή πολιτική είναι στην καρδιά όλων αυτών των θεμάτων. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε τις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα κανονισμό όπου θα καθορίζουμε τα νούμερα, την ευελιξία, τους κανόνες Χρειαζόμαστε μια διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν που θα ρυθμίζει το πώς θα διαμορφώνονται οι αιτήσεις προπολογισμοί. Και το πιο σημαντικό, η όλη δουλειά για την νομοθετική βάση συνεχίζεται. Έχουμε 17 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, τα οποία διαπραγματευόμαστε σε διαφορετικά φόρουμ. Και ξέρω ότι βουλευτές από αυτή την Επιτροπή ε, έχουν συνεδριάσεις πολλές κάθε εβδομάδα και πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου προκειμένου να καθορίσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ε, περιφερειακές πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε για την νομοθετική βάση και για το δημοσιονομικό πλαίσιο αρκετά νωρίς, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε το δρόμο για τα νέα προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να κάποια στιγμή να εφαρμοστούν κιόλα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα θυμάμαι, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις, είχαμε τελειώσει ουσιαστικά το Μάιο. Αλλά τώρα για τον προϋπολογισμό δηλαδή στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, μόλι αρχίσαμε. Άρα δεν είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Εμεί όμω, ε, ω πολιτικοί έτσι εκφύσεω είμαστε αισιόδοξοι. Και θέλω να σα πω ότι για εσά, για την περιφερειακή πολιτική, το μεγάλο τμήμα του προπολογισμού καθορίζεται στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο αναέτος και στον κανονισμό περιγράφεται χώρα προς χώρα. Δεν μπορείτε να αλλάξετε πολλά δηλαδή από χρόνο σε χρόνο στον ετήσιο προπολογισμό, αυτή στιγμή αποφασιστεί. Επομένως, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε για αυτά τα θέματα. Για τις πληρωμές έχουμε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2 από την Κομισιόν που προτείνει ότι τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσουν 11,2 δισεκατομμύρια στον προπολογισμό φέτος ε, που θα δώσει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε τους του λογαριασμούς από πέρυσι και επιπλέον θα δώσει τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που τρέχουν φέτος. Αυτό το νούμερο, το 11,2, δεν είναι τυχαίο. Είναι το ποσό που βρίσκεται στο περιθώριο. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Αν χρειαστεί να ξεπεράσουμε αυτό το ποσό, θα χρειαστούμε ομοφωνία και αποκλείεται να την έχουμε. Ακόμη και με την ειδική πλειοψηφία, και αυτή να επιτευχθεί δεν είναι καθόλου εύκολο στο Συμβούλιο, θα είναι δύσκολο να διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο ε, και επομένω ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, εμεί στην Επιτροπή Προπολογισμών. Η απογοήτευσή μας στην Επιτροπή μα είναι ότι βλέπουμε ότι το βασικό πρόβλημα με τι πληρωμέ βρίσκεται στην περιφερειακή πολιτική όπου είναι πάντα πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε πότε τελειώνουν τα προγράμματα, πότε πρέπει να πληρωθούν και βεβαίως οι πληρωμές αυξάνονται κατακόρυφα στο τέλος της περίοδου. Όλα αυτά τα ξέρετε πολύ καλά. Όταν καθυστερούμε τις πληρωμές των λογαριασμών, δεν ακούμε πολλά παράπονα από τις περιφέρειες ή τις χώρες που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρουν τα λεφτά. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη και χρειαζόμαστε τα άτομα τα οποία θα πάρουν τα λεφτά να υψώσουν το ανάστημά τους. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν. Γιατί αλλιώς πώς θα πείσουμε το Συμβούλιο ότι υπάρχει πρόβλημα αν δεν μιλάνε αυτοί που πρέπει να πάρουν τα λεφτά. Ακούμε από ερευνητέ που, που προωθούν προγράμματα στην έρευνα κτλ ότι όταν δεν πληρώνονται, ας πούμε, οι λογαριασμοί στο 1α, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να πληρώσει επιτόκια ε, για τις υπερημερίες. Αλλά αυτό δεν ισχύει καθόλου στην περιφερειακή πολιτική. Τα πράγματα είναι πιο, τα όρια είναι πιο ευέλικτα. Άρα, εσείς θα πρέπει η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής και οι υπεύθυνοι για αυτά τα προγράμματα στα κράτη-μέλη να ορθώσουν το ανάστημά τους, να μιλήσουν και να πούν ότι και για την περιφερειακή πολιτική είναι σημαντικό να πληρώνονται οι λογαριασμοί εγκαίρως. Όπως είπε και ο κύριος Σταυρακάκης, η Κομισιόν θα ετοιμάσει μια πρόταση για τον προϋπολογισμό του 14 το Μάιο. Φαντάζομαι τέλος Μαΐου θα είναι έτοιμη αυτή η πρόταση. και στην πρότασή τους θα διαμορφωθεί η απαρχία του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Υποτίθεται θα, θα είναι σαν να ανακαλύπτουν, ας πούμε, ότι συναντήθηκαν το Φεβρουάριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και αποφάσισαν. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόταση θα πρέπει να συνεχίσουμε μετά όλοι μας τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να ξανάρθω στην Επιτροπή σας καθώς θα προχωράει η διαδικασία του προϋπολογισμού για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τελευταίο σχόλιο, έτσι πιο πρακτικής φύσεως. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και από καιρούς καιρών υπάρχουν και στην Επιτροπή σας. Αν έχετε ιδέες λοιπόν, θέλω να πω, για τον τομέα αυτό, για τα πιλωτικά, έτσι θα πρέπει να τα υποβάλλετε μέχρι τέλος Μαΐου στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αξιολογούνται από την Επιτροπή και βλέπουμε αν οι ιδέες αυτές είναι κατάλληλες για πιλωτικά προγράμματα ή προπαρασκευαστικές δράσεις και αν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τα ισχύοντα προγράμματα. Αυτό είναι ένα πρακτικό που ήθελα να πω. Κατά τα άλλα, σε ευχαριστώ που με καλέσατε και περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίω και δεν, σας, ε, δεν περιμέναμε να μα ε, φτιάξετε το κέφι, αλλά βλέπουμε ότι και εσεί κατανοείτε τι είδου πρόκληση αποτελούν αυτά τα ζητήματα του προπολογισμού για την ε, Επιτροπή μας και όπως ξέρετε από όλο αυτό το ποσό τα 9 δις αφορούν την περιφερειακή πολιτική. Έχουμε λοιπόν καθυστέρηση πληρωμών όχι μόνο το 2013 αλλά κάποιες πληρωμές δεν ξέρω ποιο είναι το μερίδιο που αφορούν ε, τον, ε, το κλείσιμο του της περίοδου 2000-2006. Έχουμε εδώ τους Σούριαν, να έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση και από πλευράς εισήγηση από την Επιτροπή Προϋπολογισμών μιλώντας για αυτά τα θέματα χαιρετίζω την Άννα Γένσεν που κατάφερε το ακατόρθωτο και παρακολουθώ εδώ και δέκα χρόνια τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά ιδιαίτερα την περιφερειακή πολιτική και υπάρχει ούτε από τους πιο πεπειραμένους δεν άκουσα κάτι τέτοιο ότι μια εισηγήτρια τον Απρίλιο τα ουσιοδέστερα στοιχεία δεν μπορεί να τα γνωρίζει, λέει, γιατί δεν τα γνωστοποίησε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει παρόλα αυτά, παρόλα αυτά να υποβάλει τις προτάσεις της. Χαιρετίζω εξ του ΕΛΚ λοιπόν τις προτάσεις της εισηγήτριας. Ο κύριος Σταυρακάκης πιο πριν όλα τα προανέφερε με λίγα λόγια τα οποία μας εξέφρασε. Αυτά τα οποία μπορούν να έχουν σήμερα ιδιαίτερο βάρος. Χαιρετίζει λοιπόν το ΕΛΚ αυτά που εμπεριέχονται στο κείμενο. Δεν είναι αναγκαίο λοιπόν να έχουμε τροπολογίες και να αλλάξουμε και να δυσχεράνουμε το κείμενο περαιτέρω. Δεν χρειάζεται αυτό. Μία σκέψη θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα εδώ. Ποια είναι αυτή. Είναι το ότι η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή το θεωρεί ως ένα θέμα που έχει σημασία κλειδιού, έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα δηλαδή, για να λύσουμε τα θέματα που αφορούν την τροπολογία για τον προϋπολογισμό, τροπολογίες για τον προϋπολογισμό, διότι τα περισσότερα κονδύλια στην, περιοχή, στην πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική δαπανώνται. Επίσης, επειδή το Κοινοβούλιο αυτή την τροπολογία πολύ νωρίς θέλει να, την, ε, να εγκριθεί και να περάσει. Εμείς την καταθέσαμε λοιπόν από πλευράς μας. Υπό τις αρχικές επιθυμίες του Κοινοβουλίου όμως δεν συμπεριλαμβάνεται ότι αυτή η τροπολογία, πώς να το πω, θα πρέπει να εγκριθεί πριν πριν από τη συνέχεια και ορίμανση της συζήτησης για τα πολιετή πλαίσια, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε το έργο της. Τα χρήματα φυσικά δεν επαρκούν. Όμως, επειδή ακριβώς δεν επαρκούν τα χρήματα, αυτή τη διαδικασία δεν θέλουμε να την τροχοπεδίσουμε, δεν θέλουμε να τη σταματήσουμε. Παρακαλώ τους συναδέφους ε, και προς το συμφέρον και ενδιαφέρον του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε ώστε οι συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και να κλείσουν και τα αποτελέσματα να είναι τα ευκταία. Συγχαίρω λοιπόν τον κύριο Σταυρακάκη για το πολύ καλό κείμενο το οποίο εκπώνησε εδώ και παρακαλώ τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής να εγκρίνουν το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστούμε, η Κωνσταντσε Κρέλ, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία παρατήρηση ήθελα να κάνω για τα όσα είπε η Αν Γένσεν. Διότι ουσιαστικά και εγώ θα πίστευα, μια και στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό για το 2013 ακούσαμε ήδη ποια είναι τα ελλείμματα, οι ελλείψεις που υπάρχουν για τον προϋπολογισμό και δεν μπορούν να πληρωθούν ουσιαστικά για τις περιφέρειες υπάρχει ας το πω έτσι μεγάλη οργή για το ότι εκκρεμούν λογαριασμοί και αυτό εδώ τώρα δημιουργεί προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί κάνουμε σωστά τη δουλειά μα, λένε, και δεν μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμού του. Δεν συμβαίνει όμω αυτό. Πήρα κάποιε ειδήσει που λένε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα σχέδια και προγράμματα πολλέ φορέ επειδή δεν υπάρχουν, λέει, κονδύλια. Πληροφορήθηκα. Είναι πονηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέει δυστυχώς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, αλλά όταν υποβάλλονται κάποιοι λογαριασμοί και καταλήγουν στις Βρυξέλλες κάπου, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στιγμή δεν μπορούμε να πληρώσουμε ακόμα, χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίε ακόμα και όλα αυτά αναβάλλονται, καθυστερούν για άλλους τρει μήνες, και όλα αυτά καθυστερούν για άλλους πάλι τρει μήνε τα σχέδια και τα προγράμματα. Η πραγματική, ας το πω έτσι, ο πραγματικά φλέγον, φλέγον χαρακτήρας, ε, καυτός χαρακτήρας της κατάστασης δείχνει και τις ευθύνες των ίδιων των περιφερειών πολλές φορές. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό, αλλά να μην πληρώνονται λογαριασμοί, αυτό είναι απαράδεκτο. Ποτέ δεν νομίζω ότι κάποιος το παραδέχτηκε αυτό και ήταν κάτι δεδομένο. Στις συζητήσεις μας τα λέμε εμείς αυτά εδώ. Και ίσως αυτό ε, εκφράζεται, μια και το ε, Συμβούλιο ε, έλεγε ότι δεν αληθεύουν, δεν είναι σωστά τα ποσά για τους υπολογισμούς και ότι υπάρχουν άλλοι υπολογισμοί οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ίσως εδώ υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις και το Συμβούλιο αναφέρεται σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις και ισχυρίζεται ότι δεν είναι έλλειψη λέει πληρωμών αλλά θέμα υπολογισμών και έτσι λοιπόν εδώ ε, είναι ένας φαύλος κύκλος αυτής της υπόθεσης με τις καθυστερήσεις. Εμείς από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή πρέπει στις περιφέρειες να δούμε πραγματικά αν υπάρχουν τέτοιες μαζικές καθυστερήσεις ή όχι ώστε ελλείψεις, έλλειψη πληροφοριών ε, να μπορεί να αντιμετωπίζεται για να μην υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Είναι απαράδεκτο, είναι πραγματικά κάτι εσχρό στο σβέρκο των ε, εποφελούμενων από αυτά τα σχέδια να υπάρχουν καθυστερήσεις και προβλήματα και μετά να έχουμε και μικρές ε, πόλεις, δήμους, κοινότητες που δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιες ε, καθυστερήσεις και έχουν τεράστια προβλήματα. Πρέπει να μεριμνήσουμε, να δούμε, να συλλέξουμε πληροφορίες από τις περιφέρειες που θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμες και για τις διαπραγματεύσεις για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ. Uh, thank Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε ο Γιάνν Όλμπριχτ. Ναι, Πρόεδρε. Νομίζω δύο παρατηρήσεις πρέπει να κάνω. Η πρώτη αφορά το σημερινό πρόβλημα για τις πληρωμές. Αυτό που αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα με τις ιδιομορφίες αυτής της διαχείρισης ε, από πλευρά management που είναι διαφορετική η διαχείριση όσον αφορά για παράδειγμα θέματα έρευνας ε, και τα όσα αντιμετωπίζει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Υπάρχει τριμερή εδώ συνιστόσα είναι οι εποφελούμενοι από τα κράτη-μέλη, οι υπηρεσίε, οι οργανισμοί και οι Βρυξέλλε. Και έχουμε και τι τοπικέ αρχές και τα Υπουργεία Οικονομικών όταν έχουμε θέματα πληρωμών και Βρυξέλλε επιπλέον. Και η ένταση αυξάνεται. Εκπλήσει ότι έχετε απόλυτα δίκιο ότι η φωνή της Επιτροπής των Περιφερειών είναι αποδυναμωμένη σήμερα και αναμένουμε να μπορέσει αυτό το θέμα να το θέσει σαφέστατα η Επιτροπή των Περιφερειών. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος εδώ, ότι με ένα τόσο χαμηλό επίπεδο πληρωμών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον, η περιφερειακή πολιτική θα είναι όλο και πιο δύσκολο να υλοποιείται και να πάρει σωστές ε, σωστή μορφή. Ένας από τους τρόπους να, κρατείτε, να, κρατείτε, να κρατούνται οι πληρωμές στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο είναι να δυσχεραίνονται όλες οι διαδικασίες ώστε να υπάρχουν καθυστερήσεις. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε να υπάρχει απλούστευση. Εργαζόμαστε για να απλουστευτούν τα πράγματα. Και συζητώντας το θέμα του αποθεματικού επιδόσεων και του N συν 3 και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο αυτό που χρειαζόμαστε σαφέστατα ως μήνυμα και αυτό πρέπει να αποσταλεί από τη δική μας Επιτροπή αλλά και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι σαφής εξήγηση τι σημαίνει η απουσία όλων αυτών για την πολιτική συνοχής γιατί υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι είπαν ότι ένας μονοετής προϋπολογισμός είναι εφικτός για όλες τις πολιτικές. Άλλοι είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, είναι αδύνατο. Όμως ένα σαφές μήνυμα πρέπει να περάσει, ώστε να μπορεί να συζητήσει αυτά τα πράγματα η Επιτροπή μας. Τι σημαίνουν αυτά για την πολιτική συνοχή με τους μονοετής προϋπολογισμούς. Αν υπάρξει κατακαιρματισμός για παράδειγμα ε, σε κάποιον συνιστοσών ή καθυστέρηση ενός έτους. Θεωρητικές υποθέσεις ίσως μπορεί να φανούν αυτές. Είναι όμως σημαντικό να δούμε πώς μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε δύο συναδέλφους και από την Επιτροπή την Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και για την Διεύθυνση Δημοσιονομικών προπολογισμού. Θέλει κάποιος να παρέμβει από την Επιτροπή. Κανείς. Εσείς, παρακαλώ. Δεν έχετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ, εσείς. Thank you very much, Madam Chairman. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από την DG Regio μπορώ να επιβεβαιώσω, μπορώ πραγματικά να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν και ακούστηκαν σήμερα. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη για το σχέδιο προϋπολογισμού. Έχω κάποια στοιχεία εδώ για τις ε, διεκδικήσεις ε, ε, ετούμενων πληρωμών. 16 δις ε, αιτήσεις ήταν αυτές συνολικά που δεν πληρώθηκαν το 2012 λόγω έλλειψης δημοσιονομικών κονδυλίων και για το EADF, ε, e το Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών κάτι καταφέραμε να πληρώσουμε από όλα αυτά. Υπάρχει όμως πολύ σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά τις αιτήσει και τα κονδύλια που εκκρεμούν και πρέπει να πληρωθούν. Επιτρέψτε μου να πω, μιλήσατε πρόεδρε για το κλείσιμο του, του προγράμματος 2006. Ουσιαστικά τι βλέπουμε, έχουμε εξαντλήσει τα κονδύλια για το κλείσιμο και των προγραμμάτων και σχεδίων για το Ταμείο Συνοχής και για την, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Αν δεν υπάρχει πρόσθετος ε, συμπληρωματικός προϋπολογισμός δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε. Χρειαζόνται 1,71 δις επιπλέον. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Αν χρειάζεστε πρόσθετα στοιχεία με ευχαρίστηση να τα διαθέσω. Ολοκλήρωσα ευχαριστώ. Λοιπόν, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα μια σημαντική πρόκληση. Υπάρχει ανάγκη να πραγματικά να υψώσουμε τη φωνή μας και εμείς και να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Κοινοβούλιο. Αν δεν θέλει κάποιο από την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, Γιώργο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιάνσεν για τι πολύ χρήσιμε πληροφορίε που έδωσε στην Επιτροπή μα και όλου του συναδέλφου για την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Και Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να ληφθεί ακόμα απόφαση, εκτός και αν, αν θες να πεις κάτι. Βεβαίως. Ναι. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για τις ε, παρατηρήσεις που άκουσα και θα ήθελα κι εγώ να τονίσω τα όσα είπαν συνάδελφοι, όπως κυρία Κρέγγ είναι κρίσιμη σημασία να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσει για να ε, μάθουμε το πραγματικό μέγεθο του προβλήματο. Γιατί πράγματι υπάρχει περιθώριο ευελιξία. Ε, το έχουμε δει και σε άλλου τομεί. Ε, πρώτα από τον τομέα της έρευνας ήρθαν και μου είπαν γιατί δεν παίρνουμε τις πληρωμές για τα, για τα προγράμματά μας. Το ίδιο ερώτημα μου κάνουν ξανά και ξανά. Αυτός είναι ένας τρόπος που η Επιτροπή μπορεί να πάρει ακόμα λίγο χώρο να ανασάνει. Όμως το πρόβλημα της Επιτροπής Προπολογισμού και η θέση είναι ότι δεν πρέπει απλώς να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Είναι ένα τεχνικό θέμα και όταν υπάρχει ε, θέμα πληρωμών πρέπει να καταβάλλονται τα χρήματα. Σε πολλές περιπτώσεις ε, χρησιμοποιούμε πόρους εκεί που δεν πρέπει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και σας για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αγανάκτηση και προβληματισμό. Πρέπει να εκτιμήσουμε καλύτερα το, το μέγεθος του προβλήματο και να ε, ακουστούν και αυτές ε, οι περιπτώσεις όπου δεν καταβάλλονται πληρωμές. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Πρέπει να ληφθεί ακόμα απόφαση. Η προθεσμία ε, κατάθεση τροπολογιών 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι προτείνω εγώ και κατάλαβα ότι ο κύριος Σταυρακάκης ε, περιμένει τη συμβολή σας εν είδη τροπολογιών, ούτω ώστε να ενσωματωθούν και επιπλέον ιδέε και να επεκταθεί και η αρχική εκδοχή, η οποία βεβαίως πρέπει να είναι όσο δυνατόν βραχύτερη. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Ζαν Ζακόμπ Μπισέπ είναι μαζί μας. Ε, εντάξει, ας εξετάσουμε λοιπόν ε, την ε, ε, έκθεση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω σήμερα αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Τεχνολογία των Μεταφορών Γενικά, ε, ετοιμάζοντας αυτή τη γνωμοδότηση, εστιάστηκα κυρίως στην ιδέα ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία θα πρέπει να εξυπηρετεί την εδαφική συνοχή, ε, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υποφεληθούν και κυρίως οι διασυνοριακές περιοχές. Τόνισα την ανάγκη διάρκειας, αυτή την ανάγκη θα πρέπει να υποστηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια ε, έρευνας και καινοτομίας. Επίσης, τόνισα την εξειδίκευση. Η ιδέα της εξειδίκευσης και της έξυπνης εξειδίκευσης για να μετρήσουμε τη διάρκεια των τρόπων μεταφοράς μας είναι σημαντική για την έρευνα και την, τεχνολογία, και την καινοτομία. Μια τεχνολογία δεν είναι βιώσιμη από μόνη της. Είναι βιώσιμη μέσα σε ένα πλαίσιο. Μέσα σε ένα πλαίσιο χρήσης της και εκεί θα πρέπει να αξιολογούμε την ε, διάρκεια της. Τώρα, για να μπούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να σκεφτούμε τα ενσωματωμένα μοντέλα, της ε, τα διασυνοριακά κομμάτια μεταφορών και τις πολύτροπες μεταφορές. Αυτή είναι η προσθέμενη αξία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Επίσης, ε, μίλησα για την έννοια της διάρκειας των μεταφορών μας, θυμίζοντας οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία στις μεταφορές, θα πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τους στόχους της Ένωσης σε ό,τι αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, επικεντρώθηκα στην έννοια της εξειδίκευσης, της έξυπνης εξειδίκευσης, που πιστεύω ότι είναι μία από τις βασικές έννοιες που πρέπει να αναπτύξουμε στον τομέα αυτό. Επίσης, ε, εξήγησα γιατί οι νησιωτικές ε, ορεινές ή αεροκατοικημένες περιοχές που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα πρέπει να υποφεληθούν από μία δική τους ε, προσέγγιση. Δηλαδή, ας πούμε, σε μία ορεινή περιοχή, τα τελεφερίκ είναι πολύ πιο σημαντικά από την κατασκευή, ας πούμε, ενός σιδηροδρόμου. Η διάρκεια ε, είναι πάντα σχετική και η καινοτομία θα πρέπει συχνά να εστιάζεται σε συμπεριφορές και στη χρήση, και στη χρήση των τεχνολογιών, παρά στην ίδια την τεχνολογία. Επομένως, θα πρέπει να εξειδικεύσουμε την προσέγγισή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα διορθωτικά ταμεία και, τα, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις είναι εκ των όνου για να αναπτύξουμε την έξυπνη εξειδίκευση εφαρμοσμένη στην βιώσιμη και διαρκή κινητικότητα. Το τόνισα αυτό. Επίσης υπενθύμησα ότι οι διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να απλουστευτούν και ότι η πρόταση του συστήματος τρίνης θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τις μεταφορές. Ξέρουμε ότι αυτές οι πληροφορίες ε, δεν είναι αρκετά προσπελάσιμες από τις περιφερειακές αρχές, δεν τις ξέρουν. Ε, καταληκτικά θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζω το κείμενό μου να είναι ισορροπημένο και να είναι αποδεκτό από εσά. Φυσικά είμαι ανοιχτός σε παρατηρήσεις και σε προτάσεις τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Γιώσεφ Ματούλα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά, η Λευκή Βίβλος αναφέρεται σε μια ευρωπαϊκή περιοχή μεταφορών. Είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο στόχος. Ε, διατροπικές, ε, ολοκληρωμένες, ενσωματωμένες μεταφορές είναι μια ιδέα από την οποία πόρο απέχουμε. Λογικό είναι όμως να κοιτάμε προς το μέλλον και να βλέπουμε, να ταινίζουμε το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών. Γιατί θέλουμε ε, οι άνθρωποι και τα αγαθά στο μέλλον να, να μετακινούνται πιο εύκολα, ε, να μειώσουμε το κόστος, ε, τη χρήση της ενέργειας, ε, να είναι πιο βιώσιμες οι μεταφορές. Οι στόχοι βεβαίως είναι πολύ φιλόδοξοι. Το 96% των ευρωπαϊκών μεταφορών αυτή τη στιγμή βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα και στα παράγωγά τους. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική μεταφορών, ούτω ώστε να να αναπτύξουμε ευρωπαϊκές υποδομές που να είναι βιώσιμες. Επίσης, πρέπει να συμπληρώσουμε τους ε, ελίποντες ε, κρίκους ε, Παραδείγματο χάρη στι αεροκατοικημένε περιοχέ, στι συνοριακέ περιοχέ. Εκεί κάτι λείπει, ούτω ώστε και να βελτιώσουμε επίσης την ήπια υποδομή στις ε, μεταφορές για να αυξήσουμε την κινητικότητα, να μειώσουμε τη συμφόρηση και να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τους φορείς της, ε, του κλάδου των μεταφορών. Φυσικά θα πρέπει να υποφεληθούμε από το υπάρχον δυναμικό. Μην ξεχνάμε ότι μια έρευνα του 2008, μια επένδυση διορθώνει ο μιλητής, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ήταν, ε, η επένδυση αυτή ε, έφτασε στο ύψος των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο τομέας αυτός είναι τεράστιος, είναι πολύ μεγάλος. και επενδύει πραγματικά ο τομέας αυτό στην έρευνα και θα πρέπει να υποφεληθούμε από αυτήν την προσπάθεια. Μην ξεχνάμε τις διαφορές όμως μεταξύ των περιφερειών. Δεδομένου του κατακαιρματισμού που υπάρχει και των διαφορών, υπάρχουν πολύ διαφορετικές ιδέες, πολύ διαφορετικά προγράμματα που κυκλοφορούν και που αξίζουν της υποστήριξής μας. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, για να ανθίσουν και νέες ιδέες, να κυκλοφορήσουν νέες ιδέες. Το πρόγραμμα Ρήνου Δούναβη, ο διάδρομος αυτός, είναι ένα παράδειγμα σιδηροδρομικής μεταφοράς αγαθών σε μεγάλη απόσταση. Αν ενσωματώσουμε και του περιφερειακού φορεί, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε εταιρικέ σχέσει βιώσιμε για τι μεταφορέ, αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Και αυτό υπάρχει στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και στη στρατηγική του 2020. Σε ό,τι αφορά τι αστικέ περιοχές και τις ε, διαστικές μεταφορές, εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί Ξέρουμε πόσο χρόνο χρειάζεται να ξοδεύει κανείς, ας πούμε, στο αυτοκίνητό του κολλημένο στην, κίνηση. Ε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά ε, για επιμερισμένες μεταφορές. Να μοιράζουμε, ας πούμε, να χρησιμοποιούμε από κοινού ποδήλατα, ε, αυτοκίνητα, περισσότερους πεζόδρομους ή περισσότερους δρόμους ειδικά για, ειδικούς για, το, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε το πρόγραμμα ε, για το διαβατήριο για τα, για τα ποδήλατα στην Ευρώπη. Υπάρχουν μία σειρά από ιδέες, πρέπει να τις προωθήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να διαδώσουμε τις πληροφορίες. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά για να εντοπίσουμε τις ανάγκες. Η μερίδα, πούμε, ανοιχτών θυρών. Ε, προγράμματα βιώσιμα για τις αστικές περιοχές που συντάσσονται με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά είναι πολύ επιβοηθητικά και μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών σε τρίτες χώρες. Καταληκτικά, η έρευνα και η καινοτομία σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να εστιάσετε στα μέσα των μεταφορών, στην υποδομή και και στην αρχή της διατροπικότητας, των διατροπικών δηλαδή μεταφορών, ειδικά στις αστικές και διαστικές περιοχές. Συγχαίρω τον ε, εισηγητή και ελπίζω να συνεργαστούμε. Από... Για τους σοσιαλιστές Γιάννης Νίλσον, ευχαριστώ πρόεδρε. Από πλευρά εισηγητή έγινε καλή δουλειά με αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, πιστεύω. Είναι σημαντικό τα μέτρα, όχι μόνο να υιοθετούνται για τη δημιουργία υποδομών στην Ευρώπη, αλλά να δημιουργήσουμε και τις τεχνικές με τις οποίες θα το κάνουμε αυτό. Διότι θα χρειαστούμε υποδομές που θα είναι βιώσιμες και αηφόρες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ενιαίου πλαισίου μεταφορών. Για να διασφαλιστεί αυτό πρέπει κάποιες περιφέρειες είτε μειονεκτικές είτε εκείνες που έχουν φυσικά μειονεκτήματα δεν θα αποκλείονται. Οι υποδομές είναι συχνά το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία ανάπτυξης ε, του δυναμικού για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είχαμε χθε ένα παράδειγμα για την Σουηδία. Φανταστείτε να γίνεται αυτό με έλλειψη υποδομών ως εγχείρημα. Για να αντιληφθούμε το μη εκμεταλλευτικό εκμεταλλευόμενο από πλευρά μα δυναμικό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνικέ μεταφορών και οι λύσει κινητικότητα θα αναπτυχθούν σε περιοχέ που έχουν το δυναμικό και για την έρευνα και ανάπτυξη. Και εδώ η πολιτική συνοχή διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να υπογραμμιστεί, να τονιστεί αυτό και στη γνωμοδότησή μα. Όπω είπα στην αρχή, το σχέδιο γνωμοδότηση είναι καλό. Θα καταθέσω κάποιε τροπολογίε για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η σκιώδη όχι τώρα από πλευρά σας θέλετε να παρέμβετε ευχαριστώ πολύ πρόεδρε δεν έχω τίποτα να προσθέσω δεν έχω μεγάλα πολλά σχόλια να κάνω θέλω μόνο να τονίσω ότι ιδιαίτερα και ειδικά τα νέα κράτη-μέλη χρειάζονται βελτιώσεις όχι μόνο στις τεχνικές αλλά επίσης και υποστήριξη γενικότερα για τις υποδομές όπως προαναφέρθηκε από τον συνάδελφο Νίλσεν. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια στον συντάκτη γνωμοδότηση συζητητή. Από τους συναδέλφους της Επιτροπής υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να παρέμβει. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε για την... το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Καινοτομία και τεχνολογίες έχουν κύρια σημασία για τον τομέα μεταφορών και την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Όχι μόνο σε σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την υλοποίηση και υιοθέτηση αυτών των λύσεων και προτάσεων. Η περιφερειακή πολιτική είναι ένα σημαντικό μέσο για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Ε, επιπλέον είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους μήνες διαβουλεύσεων και συζητήσεων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στον τομέα των μεταφορών να δοθούν σημαντικά κονδύλια για την έρευνα και τον ορίζοντα 2020 υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των ε, μέτρων και των πολιτικών μεταφορών για την ενίσχυση της ε, συνεκτικότητας και συνοχής και οι τεχνολογίες για, αυτό το τμήμα είναι πολύ σημαντικό ενδυναμώνοντας ε, την Ευρώπη και δίνοντας ωφέλη για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια ευρεία προσέγγιση. Οχήματα πρέπει να δούμε που πρέπει να επιτύχουμε να γίνουν πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά. Η χρήση αυτών, η υλοποίηση του συστήματος μεταφορών, οι υποδομές πρέπει να τύχουν κινήτρων. Αυτά τα κλειδιά και η δύναμη στην καινοτομία οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ διαφορετικών πεδίων και τομέων καινοτομίας. Η ευφυής πόλης είναι μέσα στην εταιρική σχέση ευφυών πόλεων κάτι σημαντικό. Δηλαδή θέματα ενέργειας, θέματα περιβάλλοντος, θέματα μεταφορών, σημαντικά και για τα θέματα έρευνας. Περιορίζομαι στα σχόλιά μου εδώ. Ευχαριστούμε και πάλι για την υποστήριξη, για την ανάπτυξη για τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλο που να θέλει να παρέμβει. Εσείς και σε θέλετε να προσθέσετε κάτι για να ολοκληρωθεί. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, που παρενέβησαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρθηκε στις ε, πτυχές του υπερπολογισμού που σχετίζονται με, την, με τις ευφυείς μεταφορές σε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό δίκτυο και περιμένω βεβαίως με ανυπαμονησία τις ε, τροπολογίες σας και θα τις εξετάσουμε από κοινού. Ε, Ευχαριστούμε. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση για την ε, κατάθεση τροπολογιών. Προτείνω και πάλι 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Τότε λοιπόν ε, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Κλείνει αυτό το σημείο της μέσης διάταξης. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ε, Ω συνήθω θα ήθελα να ελέγξουμε το μηχάνημα. Α, έχουμε 5 λεπτά ακόμα μπροστά μας. Πρέπει να περιμένουμε. Oh, I mean, the how... Οι συντονιστές βέβαια αποφασίζουν ε, Ποια είναι η άποψή σας. Αλλά μάλλον ε, μπορεί κάποιος να έρθει ακόμα. Yeah, you cannot put it so out. I, I understand we, we, may, we have a technical pause of four minutes just. Ας κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο τεχνικό διάλειμμα 5 λεπτών και θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία στις 10. Ε, ε, ε, Συνάδελφοι, είναι 10. Ησυχία παρακαλώ. Seated. Can we check the... Ας ελέγξουμε τα μηχανήματα. Βάλτε παρακαλώ τις κάρτες σας για να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Okay, yeah, but, but if I go here, I just look here. At, uh... Να ελέγξουν όλοι οι συνάδελφοι. Δεν έχετε ψηφίσει όλοι. Αν θέλετε να ελέγξετε την κάρτα σας για να ξέρετε και αν δουλεύει. Um, Κάποιοι δεν θέλουν ε, να ψηφίσουν. It's moving all the time. Okay, we close δεν έχουν ψηφίσει όλοι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν τι ψηφοφορίε με την υιοθέτηση του σχεδίου έκθεσης ε, του Γιάννη Γκάιερ. Διακόπτη πρόεδρο, Για τι περιφερειακέ στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές. Ε, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. είναι πολύ δύσκολο να δω, γιατί πολύ λίγοι από εσάς σηκώνουν το χέρι σας. Φαντάζομαι ότι έχει υιοθετηθεί, αλλά από εδώ και πέρα παρακαλώ να υψώνετε το χέρι σας. Η ε, συμβιβαστική δύο υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 20 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ. Να ελέγξουμε εδώ, στην τροπολογία 21, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απερίφθη 16 με 18. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλους κατά Βίκτορ. Φτάνουν. Ωραία, συνεχίσουμε. Πρόταση 1 από την ΕΜΒ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πρόταση... Α, περνάμε στην συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Πρόταση 7 της ένβη. όπου έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ του πρώτου μέρους, κατά αποχές Υιοθετείτε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πρόταση 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 9 υπέρ, να ελέγξουμε την 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Και απορρίπτεται. 16 υπέρ, 24 κατά. 29, τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 2 υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείται. 47 υπέρ, τροπολογία, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε τη 47. Άρχεται, πέρας και απορρίπτεται 19 υπέρ, 23 κατά. Ψηφίζουμε τη 48 λοιπόν. Υπέρ, κατά, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε τη 48. Πέρας ψηφορίας και υιοθετείται. 23 υπέρ, 18 κατά. Πάμε στην πρόταση 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 ίσως υπερβαίνει την αρμοδιότητα της Ρέτζη. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πρόταση 5, υπέρ. Ας ελέγξουμε την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 16 με 26. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Πρόταση 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 59. Υπέρ, κατά, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ψηφίσουμε. Για την 59 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 υπέρ 19 κατά. Υιοθετείτε, <laughs> λέει η πρόεδρος. Είπα απορρίπτεται, συγγνώμη. Κάποιοι ψήφισαν διαφορετικά. Λοιπόν, υιοθετείτε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 1. τη ψηφοφορία. Υιοθετείται. 26 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά. Αποχέ. υιοθετείται. 3 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 7 υπέρ κατά ελέγχουμε την 7. Πέρας ψηφοφορίας υιοθετείται 22 υπέρ 19 κατά. 8 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε και πάλι. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Υιοθετείτε 28 υπέρ 14 κατά. 9 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Απορρίτεται. Νομίζω υιοθετείτε. Να ελέγξουμε τη 10. Πέρας. Εγκρίνεται. 27-15. Και έχουμε την τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 31 εναντί μια ψήφου εναντίον εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Περνάμε στο επόμενο Σαν Σανκέλης έκθεση. γνωμοδότηση είναι, λέγεται στην πρόεδρο. Σον Κέλλη. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Γνωμοδότηση Σον Κέλλη. Τροπολογία συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 5 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 17 υπέρ 25 ε, εναντίον. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 τώρα. Τροπολογία. Θα ψηφίσουμε τη 14. 14 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Υπέρ του πρώτου τμήματος. Θα ελέγξουμε το πρώτο τμήμα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα της 14. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 18 υπέρ 24 εναντίον. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 33 υπέρ θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 33 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα απορρίφθηκε 18 υπέρ 25 εναντίον 34 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 42 υπέρ, ένας εναντίον. Συγχαρητήρια κύριε Σον Κέλλη. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τώρα Ρίκα Μάνερ, βιοοικονομία για την Ευρώπη. Ψηφίζουμε. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει άλλη. Συμβασμός 2 λοιπόν, υπέρ. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, δεν κατέπεσε αυτή. Ωραία. Τροπολογία 4 λοιπόν τώρα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 4. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκε 18 υπέρ 24 εναντίον. Συμβιβασμός 2 ε, ψηφίσαμε, ψηφίζουμε την τροπολογία 8 τώρα, εντάξει. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Τροπολογία 9 θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία επί της 9. Πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 24 υπέρ, 17 εναντίον. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. 17 υπέρ. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 17 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 23 υπέρ 19 αντίον. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τοπολογία 19 αποσύρθηκε. Πάμε στην τοπολογία 23 υπέρ. Θα ελέγξουμε την 23 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 16 υπέρ 27 εναντίον. Πάμε στο συμβασμό 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, υπέρ του πρώτου. Θα ελέγξουμε το πρώτο τμήμα ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 18 υπέρ 26 εναντίον. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα επίσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 30 υπέρ 13 εναντίον. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελική ψήφιση τώρα, τελική ψηφοφορία. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 43 υπέρ 1 εναντίον. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια. Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία του κυρίου Βλάσακα για τον σχεδιασμό της ε, πολιτικής ε, Forward Policy Planning. Τροπολογία 1. Ξεκινάμε υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Θα ελέγξουμε την 5 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 26 υπέρ 18 εναντίον. Πάμε στον συμβασμό 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Θα ελέγξουμε την 9. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται πέρα ψηφοφορία. Εγκρίθηκε 29 υπέρ 14 εναντίον. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. 13. 13 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 14 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. Τροπολογία 17. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για αυτήν την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη τροπολογία 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ωραία. Το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα και πάλι της 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 17. Άρχεται. Αποσύρθηκε. Πολύ καλά. Χωρίς προφορική τροποποίηση. Λέτε εντάξει. Ποιος μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό. Εγώ σας ακολουθώ τυφλά. Τυφλά σας ακολούθησα. Κανείς δεν εξέφρασε αντίρρηση. Λοιπόν. Ήταν θετική η έκβαση. Υπερψηφίστηκε. Λοιπόν, πάμε στην τελική ψήφιση τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και 42 υπέρ κανείς εναντίον, δύο αποχές μόνο. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Τέλος ψηφοφοριών. Εδώ. Ο κύριος συνάδελφος είναι εδώ. Εσείς είσαστε εδώ. Εντάξει. Η κυρία Κρέλ λοιπόν. Έχουμε την ανταλλαγή από, απόψεων. Έχουμε και τους ε, εκπροσώπους. Δεν υπάρχει κάποιος που από ό,τι κατάλαβα λέει ο Μιλήτρια πρέπει πρώτα να ακούσουμε τον φιλοξενούμενο και μετά θα έχω δύο ή τρεις ερωτήσεις ε, και ίσως μπορούν να απαντηθούν στη συνέχεια αυτές. Εντάξει. Πρόεδρος, συνάδελφοι, το γεγονός ότι τελειώσαμε τις ψηφοφορίες, συνάδελφοι, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε και ότι πρέπει να έχουμε θόρυβο και φασαρία στην αίθουσα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας για την έκθεση Μόιτσα Κλέβα και Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τους παρακάτω προσκεκλημένους. Θα ήθελα να τους παρουσιάσω τους προσκεκλημένους του συναδέλφους. Έχουμε τον κύριο Ζουλιαν Ντιζόλ, συντονιστή πολιτικών από το Kirkwood Housing Europe. Έχουμε τον κύριο Μάρκο Τρίλινγκ από το uh, Ταμείο Χρηματοδότησης ε, Bankwatch Network Friends of the Earth Europe. Και έχουμε και τον κύριο Γκενάντι Κοντάγεφ uh, όσον αφορά την αηφόρο ανάπτυξη για την εκστρατεία αηφόρο ανάπτυξης. Επίσης από το Bankwatch Network. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτούς. Ε. Έχουμε συνολικά μια ώρα για την ανταλλαγή απόψεων Όσο πιο σύντομοι είσαστε, τόσο περισσότερο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων θα υπάρξει. Ο κύριο Ντιζόρ πρώτο που θα λάβει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση επίση πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα παρουσιάσω κάποιες συστάσεις από διαφορετικά σχέδια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, χρηματοδοτούνται από την ΕΦΗ ε, e, Πρωτοβουλία για την Ενέργεια και επίσης ε, με το δικό μας πρόγραμμα. Θα δείτε ότι οι συστάσεις τους βρίσκονται πολύ κοντά στις δικές σας προτάσεις ε, με αρκετές τέτοιες επικαλύψεις και θα είναι χρήσιμο αυτό για την έκθεση πρωτοβουλίας που θα συζητήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, εισαγωγικά, ως εισαγωγή, πολύ σύντομα, ησυχία στην αίθουσα. think I do want to have Thank you, thank you. Σας ευχαριστώ Θα προσπαθήσω να είμαι λοιπόν πολύ σύντομος. Μάλιστα. Προσπαθούσα να διασφαλίσω ότι θα υπάρξει ησυχία για να σας παρακολουθήσουμε. Ο μιλητής σας ευχαριστώ. Η πρώτη διαφάνεια εισαγωγικά. Γνωρίζετε ουσιαστικά τα πάντα γι' αυτό. Είναι μια εισαγωγή που όπως είπα αντανακλά την θλιβερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά την αποδοτικότητα της ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρία στοιχεία χρησιμοποιώ για αυτή την καταθλιπτική πραγματικότητα που πρέπει να απεικονίσουμε. Πρώτον, το πολύ γνωστό μονοπάτι ή οδός όσον αφορά τη μείωση της ε, ε, αποδοτικότητας ενέργειας. Και δεν βρισκόμαστε καθοδόν προς την ανταπόκριση στο στόχο με την 20% μείωση ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Αύξηση εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% δηλαδή με άλλα λόγια. Δεύτερον, μια πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας της προηγούμενης εβδομάδας που λένε ότι δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τα κλιματολογικά θέματα από το 1990. Δηλαδή το περιεχόμενο άνθρακα των ενεργειακών πόρων και εκπομπών ρήπων δεν έχει μειωθεί από το 1990 κυρίως λόγω της έντονης χρήσης ε, του άνθρακα στις αναδυόμενες χώρες, Κίνα, Ινδία, αλλά επίσης επειδή και στην Ευρώπη πρέπει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά αυτή την απεξάρτηση. Τρίτο στοιχείο, η κατάσταση όσον αφορά το πρασίνι, το, τα αέρια θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Όπως ε, αναφέρεται, έχουμε μια δυσχερή, δύσκολη κατάσταση συνολικά και ο άνθρακας ε, πραγματικά όχι μόνο δημιουργεί πολύ μικρά, μικρά, μικρές εισπράξεις ε, από τους πληστηριασμούς και τις δημοπρασίες ε, εκπομπών ρήπων, αλλά υπάρχουν και ερωτήματα για την ικανότητα των μέσων αυτών για να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη. Μετά από αυτή την εισαγωγή, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά μακροπρόθεσμα πρόκειται για το γενικότερο πλαίσιο για το κλίμα, κλιματικές αλλαγές και την ενεργειακή πολιτική που συζητώνται και από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο. Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα ο ρόλος της πολιτικής συνοχής έχει κέρια σημασία. Περνάω αμέσως στις συστάσεις για κάποια από αυτά τα θέματα που προανέφερα όσον αφορά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχή στην επόμενη μελλοντική δηλαδή περίοδο, προσεχή περίοδο. Όταν δούμε τα στοιχεία για την ε, ε, χρηματοοικονομική σύνοχη και συνεκτικότητα που είναι ένα από τα κύρια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένα συντελεστή είναι η συνέργεια που υπάρχει μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτικών, τη της πολιτικής αφενό και της πρόσφατης οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα από την άλλη. Αυτά που αναφέρθηκαν σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την εφαρμογή πολιτικών πρέπει να εντάσσονται στις ε, εταιρικές σχέσεις και για το πρασίνισμα. Συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών άρθρων όσον αφορά την οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας. Άρθρο 4 για τον οδικό χάρτη, ε, άρθρο 7 για τις υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών και για τις χρηματοοικονομικές πτυχές στο επιπλέον άρθρο και εδώ αναφέρομαι σε ένα από τα άρθρα που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να θεσπίσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κινητοποίηση επενδύσεων όσον αφορά τις δράσεις αυτές. Και γι' αυτό τον λόγο τα κράτη-μέλη πρέπει να διευκολύνουν τη δημιουργία χρηματοοικονομικών μέσων και εργαλείων. Βλέπουμε ότι η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα που απαιτεί από τα κράτη-μέλη σημαντική δέσμευση όσον αφορά και τα χρηματοοικονομικά κονδύλια και τις επενδύσεις και για την πολιτική συνοχή είναι ένα από τα μέσα, ένα από τα εργαλεία που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Παράδειγμα, κάποια από τα προγράμματα και σχέδια που προανέφερα ζητούν να δημιουργηθεί ένα κονδύλιο ενεργειακής αποδοτικότητας στο πιο κατάλληλο επίπεδο, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό. Τα κονδύλια θα πρέπει να στοχεύουν σύμφωνα με την υποχρέωση που, υπάρχουν από πλευράς, που υπάρχει από πλευράς των παρόχων. Κάποιες από τις υποχρεώσεις για τους παρόχους μπορούν να υλοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο ζητώντα από τους παρόχους να επενδύσουν, να ε, δώσουν κονδύλια σε αυτό το ταμείο. Γι' αυτό θα μπορούσε να συντονιστεί με τις δράσεις στα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό απαιτεί συζητήσει με τις διαχειριστικές αρχές των ταμείων και με τη διοίκηση, τις διοικητικές αρχές όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα. Κάποια από αυτά τα προγράμματα απαιτούν να δημιουργηθούν συντονισμένες δράσεις, concerted actions, όσον αφορά για παράδειγμα την έναν διάλογο μεταξύ των διαχειριστικών αρχών. Πώς θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές και πώς θα μπορούσαν με τον καλύτερο τρόπο να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ δύο διαφορετικών πολιτικών. Ενεργειακής αποδοτικότητας αφενός και συνοχής αφετέρου. Δεύτερος συντελεστής για την χρηματοδότηση και την συνοχή είναι η θεματολογική επικέντρωση. Thematic concentration ιδιαίτερα στους τριμερεί διαλόγους. Κάποιες από τις συστάσεις που έγιναν όσον αφορά αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην κατεύθυνση του να υποστηριχθεί η θεματολογική ε, επικέντρωση. Πρώτον γιατί θα δώσει κίνητρα από, για τι αρχές να δημιουργηθούν αυτά τα κονδύλια Energy Fund, δηλαδή για την ενεργειακή αποδοτικότητα, να συλλεγούν τέτοια κονδύλια δηλαδή. Δεύτερον, επειδή θα είναι ένα ιδανικό μέσο, ένας ιδανικός συνδυασμός με τα μέσα περιφερικής ανάπτυξης ε, που έχουμε στη διάθεσή μας θεματολογική επικέντρωση θα δώσει τα αναγκαία κονδύλια για την περιφερική στρατηγική, για την περιφερική ανάπτυξη που απαιτείται από πλευράς περιφερικής στρατηγικής. Αυτό θα δώσει κίνητρα στις δημόσιες αρχές να δουν ότι πρέπει να διασφαλιστούν τα ωφέλη των χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο οι θέσει απασχόληση και υπάρχουν μελέτε που δείχνουν ποιο είναι το δυναμικό για δημιουργία θέσεων απασχόληση με επαρκή κονδύλια στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχουν άλλε μελέτε που δείχνουν τα, συν, τα επιπρόσθετα ωφέλη. Και για τη Βόρεια Ιρλανδία, για παράδειγμα, αν συγκρίνουμε το εκτιμόμενο κόστο για την παραγωγή ενεργή ενέργειας όσον αφορά την, τον ανεφοδιασμό νοικοκυριών ε, υπάρχει συγκεκριμένο κόστος και αν εκτιμήσουμε την ετήσια εξοικονόμηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από αυτές τις δράσεις μπορεί κανείς να δει και να συναγάγει ότι όταν υπάρχουν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά την ανακαίνιση, την, ε, την ε, ανανέωση ε, στις δράσεις για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα μπορούν να εξοικονομηθούν 40 εκατομμύρια ετήσια. Βλέπουμε λοιπόν σε 10 ή 13 χρόνια μπορεί να υπάρξει μια απόσβεση του κόστους επένδυσης ε, για την ανανέωση κτηρίων και της στέγασης όσον αφορά αυτές τις δαπάνες. Ε, θα ζητούμε λοιπόν να εξεταστούν αυτές οι δυνατότητες των παραλλήλων αυτών παράπλευρων ωφελιών, co-benefits και επίση να δούμε πώς μπορούν τα κονδύλια για την ενεργειακή αποδοτικότητα να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει μια σειρά μελετών εδώ που πρόσφατα έγιναν και που δείχνουν ότι αν συγκρίνουμε την χρήση των κρατικών κονδυλίων αφενός για την αναγέννηση και ανανέωση της στέγασης, των κτηρίων δηλαδή και της μόνωσής τους, ενεργειακής μόνωσης και αν δει κανείς και συγκρίνει με την δημιουργία νέων οδών, νέων οδών στο οδικό δίκτυο, μπορεί κανείς να συναγάγει ότι υπάρχει θετικό όφελος για την επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω του ότι υπάρχει εξοικονόμηση και τα κονδύλια αυτά που εξοικονομούνται μπορούν να διατεθούν για, την συνολικότερη σφαιρική οικονομία για άλλες χρήσεις. Είναι περιορισμένο το εύρος αυτών των μελετών όμως θα πρέπει στο μέλλον να λυθούν όλο και περισσότερο υπόψη αυτά τα στοιχεία. Έχοντας τώρα υπόψη τους συντελεστές ε, η επιτυχούς υλοποίησης, ε, επιτυχούς ε, εφαρμογής. Έχουμε το θέμα της συνοχής και τώρα το θέμα της σωστής εφαρμογής και συμμόρφωσης. Είναι πρώτο σημαντικό να σχεδιαστούν λειτουργικά προγράμματα με άξονες προτεραιότητας και για την πρόσβαση. Ένα από τα συμπεράσματα αυτών των προγραμμάτων στα οποία είχαμε εμπλακεί και είναι ενδιαφέρον και για την μετεξέλιξη των πραγμάτων. Η ένταξη λοιπόν ε, αυτής της συνιστώσας ε, δεν είναι το πιο σημαντικό από όλα τα στοιχεία. Φαίνεται ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν προτεραιότητες που θα θεσπιστούν ή λειτουργικά προγράμματα που θα εστιάζονται αποκλειστικά στη χαμηλή εκπομπή ρήπων άνθρακα, ώστε να πετύχουμε την κριτική μάζα που χρειάζεται. Είναι καλύτερη αυτή δηλαδή η προσέγγιση. Είναι πιο αποτελεσματική αντί να έχουμε ένα λειτουργικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων που και αυτό στοχεύει στις φιλοδοξίες που έχουμε όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Φυσικά έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που υιοθετούμε όσον αφορά και τι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Αν θέλουμε να έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα θα πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες που πρέπει να θεσπιστούν και θεματολογικά ένα πρόγραμμα δράσης στοχοθετημένο για τις χαμηλές εκπομπές ιδιαίτερα για τα κτίρια και ε, νοικοκυριά μπορεί μόνο να πετύχει αν έχουμε και παράλληλα μέτρα τα οποία θα σχεδιάζονται σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι' αυτό όσον αφορά αυτές τις εδαφικές επενδύσεις πρέπει να εντάσσονται και σε ένα ολόκληρο πλαίσιο άλλων στρατηγικών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι πτυχές στην ε, αλληλεπίδρασή τους. Ένας άλλος ε, συντελεστής για την επιτυχή εφαρμογή είναι οι τοπικές κατηγορίες ή ομαδοποιήσεις που μπορούν να επιτευχθούν με την επικέντρωση στη στέγαση και στα νοικοκυριά, στα σπίτια. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από πλευρά πολιτική είναι το σχέδιο τη ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση. Υπερβολικά συχνά υπάρχει εντύπωση ότι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι όλο και μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και έτσι λένε θα δοθούν κίνητρα στις οικοδομικές δραστηριότητες και θα υπάρξει μια ας το πω έτσι στοχοθέτηση χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ουσιαστικά τα προγράμματα στα οποία εμπλακήκαμε δείχνουν ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες οδοί συνεργασίας μεταξύ μικρών και μικρομεσαίων ε, ε, επιχειρήσεων και όχι ανταγωνισμός μεταξύ τους, συνέργεια και συνεργασία και συντονισμός μεταξύ τους. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση πλαισίων όσον αφορά ε, τον διάλογο μέσα στον οποίο θα διαμορφώνονται οι δράσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχιτεκτόνων, εταιριών για την ανακαίνιση και ανανέωση κτηρίων, η συνεργασία αυτή είναι ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία για το μέλλον και θα εξοικονομήσει και κόστος ε, κονδύλια τελικά όσον αφορά τις δράσεις αυτές είναι ενδιαφέρον γιατί μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε τοπική υποστήριξη για δράσεις περιφερειακής ανάπτυξης, τοπικής ανάπτυξης. Μικρές τέτοιες ομαδοποιήσεις μπορούν να μετατραπούν σε χρήση, να, να οδηγήσουν σε χρήσιμα αποτελέσματα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον και για την πολιτική συνοχή μια και διευκολύνει μια διάχυση ε, γνώσεων και δράσεων ώστε να μπορέσει να πετύχει η στρατηγική που ακολουθούμε. Τούτων λεχθέντων αυτά είναι συνολικά η εικόνα. Ήθελα να σας δώσω κάποιες συστάσεις σε σχέση με αυτά τα ε, προγράμματα και σχέδια για την ενεργειακή αποδοτικότητα αφενός, αλλά και για τα προγράμματα και σχέδια ε, αστικής ανάπτυξης, ανάπτυξης ε, πόλεων. Και δείχνοντας αυτές τις τάσεις είναι κέρια σημασία να δούμε πώς ανταποκρίνονται όλα αυτά στην ίδια την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρκους Ρίλινγκ είναι ο επόμενο ομιλητή. Καλημέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να κάνω να σας ε, παρουσιαστώ. Είμαστε από την ε, τράπεζα CEB. Δουλεύουμε σε 14 χώρες στην, ε, από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. και χρησιμοποιούμε και τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης. Να σας δώσω κάποια νούμερα για το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα σας πω κάποια γενικά πράγματα και ο συναδελφός μου θα αναφερθεί σε ειδικά παραδείγματα από χώρες. Ε, η οικονομίες ενεργειακής έντασης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι χώρες ΣΥΗ έχουν τη διπλάσια ε, ενεργειακή ένταση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27. Κάποιες χώρες, η Βουλγαρία ας πούμε, ε, είχε ακόμα χειρότερες επιδόσεις και δεν βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια η ενεργειακή ένταση αυτή είναι ε, μια μεταβλητή, σύνθετη, που καλύπτει διάφορες πτυχές της οικονομίας, μεταξύ άλλων και τον τομέα της στέγασης. Τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε βραχυπρόθεσμα. Μέχρι το 2020 σημαίνει βραχυπρόθεσμα. Υπάρχουν διαφορετικά σενάρια και παρουσιάζω εδώ το σενάριο που θεωρείται ρεαλιστικό γιατί είναι η σχέση κόστους ωφέλους είναι καλή. Οικονομικά δηλαδή είναι θετικό αυτό το σενάριο. Όταν δούμε το δυναμικό εξοικονόμηση στην ε, στέγη στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 18% που μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι το 2020 με μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά ως προς το κόστος τους. Ε, για τη θέρμανση το ποσοστό είναι υψηλότερο ίσως, το ποσοστό εξοικονόμησης για, την, για τον ηλεκτρισμό και τα, τις συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020. Τώρα, αναχώρα. Βλέπουμε ότι στη Λετωνία υπάρχει ψηλότερο δυναμικό σε σχέση με τη Σλοβακία, ας πούμε, αλλά φτάνουμε σε ένα ποσοστό συνολικά 15 με 20% ποσοστό εξοικονόμησης που μπορούμε να εξοικονομήσουμε δηλαδή από τα νοικοκυριά μέχρι το 2020. Τώρα, σε τι λεφτά μετατρέπεται αυτό. Στην περίοδο 2007-2013 δόθηκαν περίπου 5,5 δις ευρώ. Έχουμε σε κίτρινο τα ιστόγραμμα το μισό ποσοστό που πάει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 και των 12. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 ε, έδωσε λίγο περισσότερα, έβαλε λίγο περισσότερα χρήματα, επένδυσε δηλαδή ε, λίγο περισσότερα χρήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα για κάποιες ε, επιμέρους χώρες. Τσεχία. Ένα δισεκατομμύριο για την ενεργειακή αποδοτικότητα, περίπου. Η ενεργειακή αποδοτικότητα στη, στα στέγη ε, έφτασε στο ανώτατο όριό της μέχρι το 2011, εκεί, στην Τσεχία. Το ίδιο και για τη Λετωνία, όπου μετά από σύντομη περίοδο ε, τα χρήματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα ξοδεύτηκαν. Γι' αυτό ξανά προβλέφθηκαν χρήματα για τον τομέα αυτό. Απορρόφηση τώρα. Υπάρχει πρόβλημα για μερικές χώρες εδώ. Όπως είπε και η Κομισιόν στην ε, στρατηγική ενδιάμεση έκθεσή της, όπου λέει ότι υπάρχει αδυναμία. Λόγω του, της αδυναμίας στην διοίκηση έχουμε χαμηλότερη απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτό ισχύει για τη Βουλγαρία και για τη Σλοβακία. Είναι καλύτερα τα πράγματα όμως στην Εστονία, Λετωνία και Λετωνία. Όπως σας είπα, ε, ε απορροφήθηκαν εντελώς αυτά τα κονδύλια για αυτές τις δύο χώρες για την ενεργειακή, κονδύλια για την ενεργειακή αποδοτικότητα πάντα. Η απορρόφηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κάποιες χώρες είναι αρκετά χαμηλή, ε, κάτω από το μέσο όρο των 27, του μέσου όρου, το μέσο όρο των 27 ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο συναδελφός μου θα σταθεί σε κάποιες επιμέρους χώρες. Ε, τις οποίες μελετά ιδιαίτερα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Κουντάρεφ. Δουλεύω ε, για το δίκτυο αυτό στη Βουλγαρία. Εκπροσωπώ ε, τους περιβαλλοντικούς ε, μη κυβερνητικούς οργανισμούς στη θεματική ομάδα που συζητάει αυτά τα θέματα να σας υπενθυμίσω ότι το 2009 έγινε μια τροπολογία του κανονισμού 1080 ε, που, είχε, που έλεγε αρχικά ότι οι χώρες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 2% των κονδυλίων ε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή αποδοτικότητα στη στέγη. Αυτό το ποσοστό έφτασε στο 4% με τροποποίηση. Ε, συν ένα επιπλέον ποσοστό που μπορεί να βοηθήσει και αυτό για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα σπίτια. Πόσες χώρες ε, επωφελήθηκαν από αυτήν την τροπολογία? Αυτό είναι το ερώτημα, θα το δούμε σήμερα. Είναι σημαντικό το τμήμα των συμπερασμάτων μας, γι' αυτό σας υπενθύμισα την τροπολογία του κανονισμού. Δουλεύω στη Βουλγαρία, όπως σας είπα στην αρχή, και η κατάσταση που βλέπουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα σπίτια είναι η εξή. Τα προγράμματα που υποστήθεται ότι υποστήριζαν την ενεργειακή αποδοτικότητα ξεκίνησαν μόνο μόλις το καλοκαίρι του 2012. Δηλαδή 1,5 χρόνο πριν το τέλος της περίοδου προγραμματισμού. Η χώρα ποτέ δεν επωφελήθηκε από την τροπολογία, μόνο 32 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα σπίτια, συν 8 εκατομμύρια για την κατασκευή εργατικών ε, κατοικιών που ε, εμπεριέχουν κάποια τέτοια μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας. Είμαστε σε δύσκολη θέση στη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων, γιατί ε, υπάρχει ένα θέμα ε, ιδιοκτησίας. Μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, παλιές πολυκατοικίες με 50 διαμερίσματα. Ο καθένα έχει το δικό του διαμέρισμα, διαφορετική ιδιοκτησία. Υπάρχει πρόβλημα και με την εθνική νομοθεσία, αλλά βάζει τροχοπέδι στην υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακή αποδοτικότητα Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων είναι ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδοτούν το 50% ε, τέτοιων μέτρων. Αλλά το άλλο 50% πρέπει να το δώσει ο κόσμο. Δεν, το έχει όμω. Ε, ποια είναι η επιλογή λοιπόν, δάνειο την τράπεζα. Πολλές από τις, δάνει, από τις ε, οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα δεν μπορούν να πάρουν τέτοιο δάνειο, δεν έχουν την κάλυψη. Δεν είναι φερέγγι απέναντι στην τράπεζα. Επομένως, πιστεύουμε ότι κάποιο επιπλέον εργαλείο θα πρέπει να είναι στη διάθεσή τους, δηλαδή κάποια διαχείριση, κάποιο πρόγραμμα, κάποια κονδύλια που τα διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές ή κάποιες ΜΚΟ. Επίσης, ρωτήσαμε τους συναδέλφους μας από άλλες χώρες, από το δίκτυο όπου είναι ενεργή, ενεργό το δικτύο, η τράπεζά μας. Παράδειγμα στο χάρη στην ε, Τσεχία. Υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα πρασινίσματος που προβλέπει χρηματοδότηση για τα σπίτια. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, ένα σχήμα που χρηματοδοτείται από το ETS, κάνει μια καλή δουλειά Υπάρχει και υποστήριξη χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ε, η ζήτηση είναι σοβαρή, τα αποτελέσματα είναι καλά. Για τα δημόσια κτίρια, η χώρα ε, εξάντλησε τη χρηματοδότηση του 2011. Δόθηκαν επιπλέον κονδύλια, λοιπόν, στην Τσεχία. Στην Εστονία τώρα. Τελείως αντίθετη η προσέγγιση σε σχέση με την Τσεχία. Έχουμε εδώ. Ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια υποστήριξαν τα, τα, τα, τα, τα τις επενδύσεις στα σπίτια. Είχαμε πάνω από 500 προγράμματα στην Εστονία. Ε, συμμετείχαν διάφορες οργανώσεις ε, ιδιοκτητών ε, εκεί. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά καλά. 45% εξοικονόμηση ενέργειας περίπου, αλλά οι συνάδελφοι έχουν επιφυλάξεις γιατί οι δείκτες θα πρέπει πραγματικά να μετράνε την εξοικονόμηση στα κτίρια. Υπάρχει πρόβλημα με τους δείκτες. Ουγγαρία. Ε, ήθελε να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά ταμεία για να υποστηρίξει την ενεργειακή αποδοτικότητα στα σπίτια, στην κατοικία, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν συνέβη λόγω της οικονομικής κρίσης. Η χώρα δεν μπορούσε να υποστηρίξει και να προβεί σε εθνική συγχρηματοδότηση για τα μέτρα και προγράμματα και τα μέτρα ε, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν ανεστάλησαν πριν από δύο χρόνια και δεν προχώρησαν λοιπόν, δεν υλοποιήθηκαν. Στη Λετωνία ε, ξεκαθαρίστηκε και από την παρουσίαση του Μάρκου ήδη ότι ξεκίνησε καλά η Λετωνία υποστηρίζοντας μέτρα για την κατοικία στην αρχή της περίοδου προγραμματισμού, αλλά επειδή ξεκίνησε πολύ νωρίς, μπόρεσε να αναπτυχθεί, να επιταχύνει και να αναπτύξει ε, μια πολύ έντονη ζήτηση για την τέτοια μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στα σπίτια. Εξάντλησε τα κονδύλια πριν από κάνα δύο χρόνια και εποφελήθηκε από την τροπολογία του κονισμού το 2009. Από το 2% λοιπόν από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ανάπτυξης έφτασε στο 3% χάρη στην τροπολογία, στην Πολωνία. Δεν υποστηριζόταν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ε, η κατοικία. Είχε μια μικρή, ένα μικρό φάκελο σε σχέση με το συνολικό ποσό. Ε, η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη για τα δημόσια κτίρια και οι συνάδελφοι μου έδειξαν ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια. Στη Σλοβακία. Αυτό που μας είπαν οι συνάδελφοι είναι ότι καθορίστηκαν σωστοί δείκτες ε, και μιλούσαν για τις περιοχές ή μάλλον για την ε, έκταση που, ήταν, που είχε μόνωση. Ήταν καλύτερος ο δείκτης. Ε, δεν χρησιμοποίησε και δεν εφάρμοσε τον Τζέσικα. Άρα χάθηκαν ευκαιρίες, είπαν οι συνάδελφοι, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εργατικές κατοικίες στη χώρα αυτή. Οι συνάδελφοι μου προσπάθησαν να καταλήξουν σε κάποιες συστάσεις. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό και σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις στα πλαίσια του διαλόγου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει φιλοδοξία για τα, για τα ποσά που θα διατεθούν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και το 15% των ποσών θα πρέπει να πάνε σε μέτρα ε, και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να τεθούν πολύ γρήγορα, το συντομότερο δυνατόν. Γιατί, όπως σας είπαμε, αυτή η τροπολογία είχε... Όπως αυτή η τροπολογία, εάν ε, δεν αλλάζουμε, δεν τροποποιούμε τους κανονισμούς στην αρχή της περίοδου και το κάνουμε μέσα, στο μέσο της περίοδου, τα αποτέλεσμα είναι χειρότερα. Ε, ελπίζουμε επίσης οι ευρωβουλευτές να περάσουν το μήνυμα στις χώρες τους. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει το ανώτατο όριο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς μέχρι τόσο του ποσού του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι χώρες μπορεί να είναι πολύ πιο φιλόδοξες στον τρόπο που ξοδεύουν τα χρήματα για την αύξηση της ενεργειακής επιδοτικότητας στα κτίρια. Επίσης, θέλουμε να είναι φιλόδοξα τα προγράμματα ε, και θέλουμε να υπάρχουν και μέτρα ε, διόρθωσης των προβλημάτων διαρροής της ενέργειας και εκ των υστέρων στα κτίρια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κατασκευαστούν. Επίσης, οι εργατικές κατοικίες χρειάζονται τέτοια εργαλεία. Μιλάμε για χρήματα που δεν περνάνε μέσα από τράπεζες. Προτιμησιακή μεταχείριση για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και που είναι φτωχές ή που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ένδυας. Στην Βουλγαρία παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε αργά, φτάσαμε σε επιχορήγηση μέχρι ε, και 75% ε, για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότητας ενέργειας. Και οι φτωχές οικογένειες θα υποστηριχθούν ε, κατά 100% χάρη στην συγχρηματοδότηση από την εθνική χρηματοδότηση του υπόλοιπου 25%. Επίσης, ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται ότι τα προγράμματα αυτά είναι δικά του όταν ε, τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε επίπεδο χώρας θα πρέπει ο κόσμος να εμπλέκεται. Γιατί αφορά τη δική τους ε, κατοικία, το σπίτι τους. Και θα πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται ότι εμπλέκεται στο πρόγραμμα αυτό, τι εφαρμόζεται, σε αυτό που εφαρμόζεται, στο γιατί εφαρμόζεται, ε, στο γιατί το λένε οι εμπειρογνώμονες αυτό ας πούμε και δεν προτείνουν κάτι άλλο πιο ακριβό ή πιο φθηνό κτλ. Πρέπει να να εμπλέκεται και να ξέρει τι παίζει. Επίσης, ε, θα πρέπει να καθορίζονται σωστοί δείκτες, το είπαμε ήδη, θα πρέπει να δείχνουμε ότι έγινε τόση εξοικονόμηση, αξιόπιστη. Και αυτό μπορεί να χρησιμεύσει και ως κίνητρο. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αυτά καθεαυτά, τα προγράμματα δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στα ελάχιστα όρια που θέτουν ας πούμε, οι χώρες. Θα πρέπει όπου γίνεται να είναι και πιο φιλόδοξα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όσον νουπο, θα ετοιμάσει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Επομένως, πρέπει να είναι και τα προγράμματα τα ίδια πιο φιλόδοξα. Και τελευταία και σημαντική σύστασή μας είναι ότι υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης των ευρωπαϊκών ταμείων και κονδυλίων θα πρέπει να δίδονται σε περίπλοκα προγράμματα που είναι πολύ φιλόδοξα και, εξασφαλίζουν και εξοικονομούν υψηλό ποσοστό ενέργειας. Και σε όλες τις περιπτώσεις που τα προγράμματα ε, ξεπέρνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτουν οι χώρες για τον εαυτό τους. Ευχαριστώ. Η Κωνσταντσε Κρέλ, παρακαλώ. Κανονικά δεν επεφημούμε ούτε χειροκροτούμε. Κάποιοι θα ήθελαν ίσως να το κάνουν, αλλά όχι εντάξει σε σχέση με τόσα όσα είπατε. Η Κωνσταντσε Κρέλ, ευχαριστώ Ντανούτα. Τώρα παρεμβαίνω εξ ονόματος ε, της εισηγήτριας. Ε. Δεν μπορεί να παραστεί. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις η κυρία Μόιτσα Κλέβα Κέκους στην εκλογική της περιφέρεια. Μου ζήτησε εμένα λοιπόν να παρουσιάσω κάποια θέματα και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα, θέλει τα μέτρα για την προαγωγή αποδοτικότητας ενέργειας για το μέλλον να πει ότι είναι μια συμφωνημένη οδός για το πλαίσιο και της πολιτικής συνοχής. Οι επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα μπορούν να διασφαλίσουν και να δημιουργήσουν τοπικά θέσεις απασχόλησης μέσω ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και δημιουργούν μια κατάσταση win-win, αμοιβαία επωφελή στην καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Ωστόσο όμως, πρέπει για να επιτευχθούν τα θετικά μέτρα από αυτή την επένδυση να πούμε ότι η πρόσφατη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εν μέρει άσκησε επικρίσεις για τη χρήση των κονδυλίων όσον αφορά αυτή την πτυχή. Είπε ότι επιλεγμένα προγράμματα σε σχέση με το κόστος τους πρέπει να επιτηρούνται. Αυστηρότερα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επιλογή τέτοιων προγραμμάτων όσον αφορά την χρηματοδότηση για ενεργειακή αποδοτικότητα και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο των κρατών μελών. Θα ήθελα να ακούσει τα σχόλιά σας η κυρία εισηγήτρια Κλέβα και και να δει πώς θα ανταποκριθείτε, θα αντιδράσετε στις συστάσεις της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Ποιες είναι οι δικές σας συστάσεις όσον αφορά τα προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας ως προς αυτά. Δεύτερο σημείο που θέλει να αναφέρει η κυρία Κλέβα Κέκους. Στην έκθεσή της μία από τις κύριες συστάσεις είναι να προαγάγουμε την χρήση καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέτρων και εργαλείων σε αυτό το πεδίο. Η ευφυής καινοτόμος χρηματοδότηση και στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θετική πορεία, ως καταλήτης για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ως προς αυτά θα ήθελα να ακούσει ποια θα ήταν η δική σας άποψη όσον αφορά την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων ως προς αυτό. Και πιο συγκεκριμένα, πώς θα αξιολογούσατε, για παράδειγμα, από πλευρά των κρατών μελών την δυνατότητα να υπάρξει ε, προσαρμογή του επίπεδου συγχρηματοδότησης με βάση αυτά τα στοιχεία. Αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω μια-δύο παρατηρήσεις δικές μου αυτή τη φορά. Θα έλεγα δεν είναι μόνο δυνατόν να μιλήσουμε για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στην κοινωνική στέγαση, στα κοινωνικά διαμερίσματα και νοικοκυριά. Να πάμε πιο πέρα. Μέτρα αποδοτικότητας, ενεργειακής αποδοτικότητας και για τα δημόσια κτίρια ή γενικότερα για το, τη γενικότερη στέγαση, γενικότερα. Για παράδειγμα, τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ε, χρήση ενεργειακών πόρων και αυτό πρέπει να είναι μέλος, μέρος της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας για το μέλλον. Όχι να συζητούμε μόνο να δοθούν ενισχύσεις, αλλά και να δούμε και νέα χρηματοοικονομικά μέτρα ως προς αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Καθότι γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο από πλευράς του ενέκρινε την έκθεση για την εκπομπή διοξιδίων του άνθρακα και την, ε, την επανέπεμψε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την εμπορία ρήπων την προηγούμενη εβδομάδα και όλα το αποφασίσαμε αυτό. Οι τιμές των πιστοποιητικών ρήπων έχουν μειωθεί, έχουν συρρυκνωθεί το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα πρέπει να εξεταστεί μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ως τμήμα της ε, συνολικότερη συζήτησης. Ίσως εδώ θα μπορούσαν να γίνουν κάποια σχόλια λοιπόν και από πλευρά σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Θα πάρουμε τους αγορητές, έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ο κύριος Όλμπριχτ τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια αρκετά στοιχεία τα οποία αναφέρονται από τους ε, δύο μιλητές. Πρώτον, η αλλαγή του κανονισμού το 2009 και οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής. Το συζητήσαμε αρκετές φορές και είπαμε ότι η αλλαγή της επιλεκτικότητας και του εύρους δράσης ε, κατά τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών δεν είναι η σωστή πορεία, δεν είναι το σωστό μέσο. Το αποτέλεσμα δεν ήταν εντυπωσιακό, επειδή πραγματικά τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης διανέμονται και αυτή η πρόταση απαιτούσε αλλαγή προγραμματισμού και μεταφορά κονδυλίων όσον αφορά και την ενεργειακή αποδοτικότητα ε, κτηρίων και γι' αυτό από το 4% στο 3% που θεωρητικά μπορεί να είναι ενδιαφέρον αλλά στην πρακτική εφαρμογή δεν δίνει και μεγάλα αποτελέσματα. Και σε σχέση με, τα, με την επόμενη περίοδο 2014-2020 ε, θα έχουμε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Τώρα έχουμε διαπραγματεύσεις ε, για τις επενδυτικές προτεραιότητες, investment priorities. Αυτό συνδέεται με την θεματολογική προτεραιότητα 4, χαμηλές εκπομπές ε, άνθρακα, ενεργειακή αποδοτικότητα, παρότι δεν είναι ακριβώς τα ίδια αυτά τα δύο. Τώρα συζητάμε το εύρος των δράσεων του Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης και τα θέματα επιλεκτικότητας πάσης φύσεως κτίρια τώρα εντάσσονται δημόσια κτίρια, δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και δημόσια στέγασης και κρατική στέγασης. Αυτό προβλέπεται από τον νέο κανονισμό. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω εδώ κάτι, ότι θα έχουμε για κάποιο διάστημα συζητούμε το ελάχιστο επίπεδο όσον αφορά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ιστερότερα υπό εξέταση, αλλά πρέπει να δούμε την μείωση του ελάχιστου. Και το θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε, ίσως δεν το σημείωσα, ότι το Ταμείο Συνοχής και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις του. Και θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτηρίων. Αυτό είναι κάτι το καινούριο. Οι αντιδράσει των κρατών μελών είναι διαφορετικέ από κράτο σε κράτο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει ένα καλό σύστημα, θετικό σύστημα για κτίρια και ενεργειακή αποδοτικότητα. Δεν χρειάζονται ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ για αυτή τη δράση. Αφήνω ανοιχτό το ερώτημα. Πρέπει να απαντηθεί και να επιληθεί, ιδιαίτερα διοργανώνοντας ε, και την σύνοδο για την ε, ανάπτυξη των δράσεων στις επενδύσεις ε, όσον αφορά την κρατική παρέμβαση για τη στέγαση, την ιδιωτική στέγαση για παράδειγμα και τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων, κρατικής υποστήριξης, διότι θα έχουμε και επενδύσεις ε, εδώ δημοσίων κρατικών κονδυλίων σε ιδιωτική στέγαση. Δεν είναι σαφή τα πράγματα για την επιλεκτικότητα πώς συνδέονται. Τελική παρατήρηση που δεν συνδέεται με το θέμα της στέγασης. Να μην ξεχνάμε ότι οι ευρύτερε ε, δράσεις ε, που ακολουθούνται από τη Σύνοδο Δημάρχων. Η Σύνοδος Δημάρχων υπέγραψε ένα είδους ε, σύμβασης όπου υπόσχονται να προετοιμάσουν τα προγράμματα τα ενεργειακά για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά τα επόμενα χρόνια δήλωσαν ότι θα προετοιμάσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτό, χειροπιαστό πρόγραμμα. Και τα κονδύλια του Ταμείου Ελένα χρησιμοποιούνται ως προς αυτό το στόχο. Το θέμα είναι που τίθεται για την πολιτική συνοχής. Ποια συνέχεια θα δοθεί μετά από αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με την Σύνοδο Δημάρχων. Αν σε μια πόλη κάνουν μεγάλη προσπάθεια και προετοιμάζουν έτσι, ας το πω έτσι, το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας, θα έπρεπε να ακολουθούν μια ταχεία διεργασία, fast track για την πολιτική συνοχή. Αν όχι, θα είναι μόνο συμβολικής αξίας και ουσιαστικά άχρηστη, περιττή αυτή η δράση. Η πρότασή μου είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μία οδό, μία, έναν τρόπο, ίσως από πλευράς εφαρμογή των νομικών αυτών συντελεστών και στοιχείων, να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα ενέργεια που εκπονούνται από τη Σύνοδο των Δημάρχων όταν υπάρχει ένα τέτοιο κονδύλιο ε, που δημιουργείται να είναι πιο συμπληρωματικού χαρακτήρα στο μέλλον η μία δράση με την άλλη και να αλλοσυμπληρώνονται. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα πρόβλημα. Αν θέλουμε να αφήσουμε πέντε λεπτά στο τέλος της συζήτησης για να παρέμβουν οι φιλοξενούμενοι μας, τότε έχουμε περίπου δύο λεπτά όλα και όλα. Δηλαδή, Λάμπερ, Φαν ε, ε, Νίστερ Ρόι, Αγκουράκης, Μπουστινάρο, κλείνουμε εδώ τον κατάλογο. Αν μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις παρεμβάσεις των φιλοξενουμένων να απαντήσουν τις παρεμβάσεις. Έχουν άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις και θα πρέπει να αποχωρήσουν. Να είστε σύντομοι. Μαντέλη, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του ε, συναδέλφου που παρενέβησαν. Πρέπει εδώ πέρα να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Επειδή η ενεργειακή κατάσταση σήμερα, όπω ε, αναφέρατε, είναι δύσκολη ε, και βάσει του ενεργειακού μα μοντέλου έχουμε πολύ μεγάλε εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα και αυτό δεν είναι καλό για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντο. Είπατε ότι σήμερα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργεια αλλά υπάρχει ένα τριπλό διακύβευμα, οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση άνθρακα. Γιατί ε, το, το μερίδιο του πετρελαίου, του, του αερίου ε, και του άνθρακα μειώνεται η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο τη κοινωνία μας, το βλέπουμε σε, όλες, σε όλους τους τομείς, στην ενέργεια, στι υποδομέ, αλλά ο βασικός ε, τομέας όπου θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει η δέσμευση της Ευρώπης και εγώ συγγράφω ε, μία ε, έκθεση που θα ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα, είναι ο τομέας της εστέγασης. Βασική επίπτωση είναι, όπως αναφέρετε κι εσείς, αυτό το περιθώριο του 4% που είναι ένα πραγματικό σημείο μόχλευσης ε, ε, όπου όμως υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση γιατί δεν υπάρχει στήριξη, ε, οικονομικός μηχανισμός ούτως ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα μέσα και ε, να έχουμε τέτοια προγράμματα ενεργειακής καινοτομία. Και βρήκατε πραγματικά το επίκεντρο του προβλήματος στη στέγαση. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα. Ότι η χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων ε, ενεργειακής ε, αποδοτικότητας Εκεί το ζήτημα λοιπόν είναι το πού βρίσκουμε τα χρήματα, πού βρίσκουμε χρηματοδότηση για να υπάρχουν τέτοιες θερμικές ανακαινήσεις σε μεγάλη κλίμακα. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα πραγματικό ε, ταμείο ε, σε, συνεργασία με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να υπάρχουν πραγματικές επενδύσεις και σε αυτή την περίπτωση όλοι κερδίζουν. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε εάν παράλληλα δεν δώσουμε και τα εργαλεία τις, και ευκαιρίες απασχόλησης. Χρειάζεται επαγγελματική κατάρτιση, αξιοποίηση νέων οδών. Δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Θα πρέπει πραγματικά να προσαρμοστούμε και να προσαρμόσουμε και τους ε, εργαζομένους αυτά, αυτές τις νέες θέσεις εργασίας. Και τέλος έχουμε και αυτή την ε, οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και έτσι καλούνται τα κράτη-μέλη να σεβαστούν αυτό το όριο του 3% της ανακαίνησης για τα δημόσια κτίρια. Όμως ε, δεν ε, θα κάνουμε εκεί τη μεγάλη, αλλά στη στέγαση, τα παλιά κτίρια. Εκεί υπάρχει πραγματική αξία να επενδύσουμε. Και όπως είπε και ο κύριος Αλμπρίχτ, ναι, πρέπει να ζητήσουμε από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να επενδύσει ε, και στα δημοσιακτήρια αλλά και στην ε, κοινωνική στέγαση. Εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί ε, χρηματοδότησης και ποιε είναι οι περιφερειακέ πτυχέ που μπορούμε να εξετάσουμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα. Να υπάρχουν επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο για τη θερμική ανακαίνιση. Εκεί έγκυται η δυναμική του τομέα τη στέγασης. Αναφέρθηκε κάτι σημαντικό προηγουμένω. Πολύ συχνά όταν μιλάμε για θερμική τέτοια ανακαίνιση ε, ξεχνάμε την ε, ενεργειακή επισφάλεια που έχει άμεση επίπτωση στην αγοραστική ε, δύναμη των κατοίκων. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και τον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της ενεργειακής μετάβασης. Και η σύνδεση που, είπα, που αναφέρατε και στις είναι ε, η σύνδεση μεταξύ της υγείας και της ενεργειακής ασφάλειας. Και κλείνω εδώ. Εγώ ζητώ λοιπόν από τους ε, να μας πούν εάν θεωρείτε ότι σήμερα έχει έρθει η ώρα να φροντίσουμε ούτως ώστε η Ευρώπη να αξιοποιήσει και να, θεσπίσει ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα μπορέσει να αναλάβει τέτοια, ε, τέτοιες επενδύσεις και πώς θεωρείτε ότι πρέπει να συσταθεί αυτός ο νέος χρηματοδοτικός οργανισμός. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την αξιοποίηση του Τζέσικα και των άλλων μέσων. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Απλώ δεν ε, θα μπορέσω να δώσω το λόγο στου συναδέλφου, γιατί μιλήσατε για πάνω από 5 λεπτά και τώρα έχουμε 12 λεπτά για τα υπόλοιπα. Λάμπερτ. Ένα λεπτό μόνο. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που ήρθαν εδώ ε, οι εκπρόσωποι αυτοί γιατί εστιάζεται και στην έκθεση Κρέμπα. Είπαμε και στο έλκο ότι πρέπει να είναι το βασικό ε, σημείο συζήτησης η ενεργική απόδοση. Δεύτερον, πολλά μπορούν να αλλάξουν, όμως έχουμε τα μέσα. Όμως, κατά την προετοιμασία των συμβάσεων εταιρική σχέση ε, στα κράτη-μέλη. Τι συμβαίνει, πρέπει να ξεκινήσει του χρόνου, την 1η Ιανουαρίου. Βρίσκεται στο πρόγραμμα κάθε χώρα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράση συνεργειακή αποδοτικότητα στα μέσα του έτου. Τι συμβαίνει με αυτό, Γιατί δεν αξιοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεύτερον, το ΕΛΚ δεν θέλει να φέρει νέα στοιχεία, νέες υποχρεώσεις. Ζητούμε μεγαλύτερη ευελιξία. Όμως να καταγραφούν πολύ συγκεκριμένα σε αυτές τις συμβάσεις εταιρική σχέσης και στα σχέδια ε, δράσης. Μπορούν να υπάρχουν διαφορές ε, στα κρατημέλη βεβαίως, αλλά μιλάμε μόνο για τις χώρε σύγκληση και συνοχή όμω πώ έχει η κατάσταση στι υπόλοιπε χώρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σον Κέλλη. Ναι, και εγώ πολύ σύντομα. Ήταν πολύ σημαντικό που το πρώτο που ακούσαμε ήταν η πρόοδο προ τι καθαρέ ενέργειε που έχει ξεκινήσει από το 1990. Βέβαια, δεν είναι πολύ το αυτό. Μετά όμω οι ομιλητέ είπαν κατά πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, πράγματι είχαν ε, λογικά επιχειρήματα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ροπή προς την αναβολή της ε, δράσης με το να έχουμε μακρο, μακροπρόθεσμους στόχους. Όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να δράσουμε τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Το ζήτημα της στέγασης. Υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα εδώ ο κόσμος είναι έτοιμος αν τους δώσουμε τα μέσα και τα εργαλεία. Βεβαίω, ε, το μερίδιο της χρηματοδότησης συνοχής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, αλλά για να έχουμε νέα χρηματοδοτικά μέσα, καλή ιδέα θα πρέπει να τη διερευνήσουμε. Κάτι που θέλουμε να κάνουμε στην Ιρλανδία είναι το λεγόμενο pay as you save, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει κόστος για τον ιδιοκτήτη και μετά να δούμε ότι αν έχει γίνει σωστά η δουλειά, τότε υπάρχει εξοικονόμηση. Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό όμως, κύριε Πρόεδρε, για την επαγγελματική κατάρτιση. Πολλοί καουμπόιδες έχουν ε, μπει σε αυτή την ε, κατάσταση και θα πρέπει επιτέλους να εξολογήσουμε σωστά την κατάσταση, να υπάρχει σωστή κατάρτιση και παρακολούθηση. Και τέλος, για τη Βόρεια Ιρλανδία που είχαμε εξοικονόμηση 40 εκατομμυρίων ε, μετά από αυτά τα μέτρα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο, γιατί ότι, βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν μόνο ωφέλη περιβαλλοντικά, αλλά και για τον πληθυσμό. Όσο περισσότερα κάνουμε και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριο Σαγκουράκης. Ευχαριστώ. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις να κάνω. Καταρχήν η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Τρίλινγκ. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι στο χρονικό διάστημα 7-13 δαπανήθηκαν 5,5 δις για έργα ε, ενεργειακής απόδοσης. Ε, υπάρχει κάποιο στοιχείο που να μας λέει πόσο αυξήθηκε ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης για αυτό το ποσό. Δεν το συγκράτησα. Το δεύτερο είναι ε, τρεις ερωτήσεις για τον κύριο Κοντάρεφ. Ε, ο κύριος Κοντάρεφ μας είπε ότι στην Εστονία δεν ήταν καλοί οι δείκτες. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει ποιοι θα ήταν οι καλοί δείκτες. Δηλαδή ποιοι θα έπρεπε να είναι οι δείκτες ώστε να θεωρήσουμε ότι ήταν καλοί. Δεύτερη ερώτηση, εάν ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης στις μελέτες που κάνει ανεβαίνει με το χρόνο ή μειώνεται. Γιατί φαντάζομαι όταν κάνεις μια επένδυση στην αρχή είναι σε ένα δεσμένο επίπεδο, με την πάροδο του χρόνου τι γίνεται, ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Και τρίτο, όσον αφορά τη Βουλγαρία, έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα και στην Ελλάδα. Τώρα, χαριτολογώντας από το εξή. Είναι τραγικό, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Δυστυχώ φάνηκε ότι ο καλύτερο τρόπο ενεργειακή εξοικονόμηση είναι η καπιταλιστική κρίση. Στην Ελλάδα η κατανάλωση ενέργειας έχει πέσει 30% στα νοικοκυριά Πολύ απλά διότι είναι πολύ ακριβή ενέργεια, είναι πολύ ακριβή και το πετρέλαιο και η ηλεκτρική ενέργεια και έχουμε την καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Στη Βουλγαρία ξέρω ότι έπεσε η κυβέρνηση λόγω των τιμών, των πολύ ψηλών τιμών στη, στο θέμα της ε, ενέργειας. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί και τέλος, γιατί δεν, ε, οι αξιότιμοι συγητές μας δεν επικεντρώθηκαν λίγο περισσότερο στα δημόσια κτίρια, σε επιχειρήσεις, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Ευχαριστώ. Thank uh, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω το θεμελιώδες ερώτημα πρέπει να διατυπώσουμε. Τι θέλουμε να πετύχουμε με την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε τις περιφέρειες πιο ανταγωνιστικές. Θέλουμε να έχουμε πολιτική κατά των κλιματολογικών αλλαγών. Αυτή η θεμελιώδης ερώτηση πρέπει να τεθεί ως ερώτημα. Και επικεντρωνόμενη σε σχέση με τα σπίτια της στέγαση είτε είναι κρατικού είτε ιδιωτικού χαρακτήρα θέτω το ερώτημα γιατί μια περιφέρεια με καλά μονομένα ε, κτίρια μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική από άλλες. Αυτό το ερώτημα πρέπει να θέσουμε για να το βρούμε την απάντηση. Διότι σε σχέση με την πολιτική συνοχή το πρόβλημα είναι όταν έχουμε πράγματα τα οποία εντάσσονται στην ενεργειακή αποδοτικότητα όπως ε, την μόνωση βοηθούμε μόνο με μια συγκεκριμένη τιμή να είναι πιο ανταγωνιστικές οι περιφέρειες σε σχέση με τις επενδύσεις που θα γίνονται σε έναν τομέα που θα έχουν πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα στις επιπτώσεις τους. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το σκηνικό με την οδηγία ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι ο μόνος από τους τρεις στόχους που δεν θα επιτευχθεί από ό,τι φαίνεται. Κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση και τα κράτη-μέλη δεν ήταν καν πρόθυμα την ενεργειακή αποδοτικότητα ως δεσμευτικό στόχο να την εντάξουν και με πολλά δεσμευτικά μέτρα. Να υπενθυμίσω ότι η ίδια η οδηγία ενεργειακής απόδοσης μόνο τον ε, ουσιώδη ε, τομέα θίγει και όχι τον ε, ιδιωτικό, τον κρατικό και όχι τον ιδιωτικό. Τώρα εντάσσονται αυτά στην πολιτική συνοχής Πρέπει να δημιουργήσουμε τις σωστές παραμέτρους ε, και το ζήτησε αυτό και το ελεγκτικό συνέδριο. Και στην τελική περίπτωση πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο σε σχέση με τη θέρμανση κτηρίων για παράδειγμα. Και μετά βλέπουμε ότι ε, κάνουμε συγκεκριμένα λόγο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αν δεν ξεχωρίσουμε και δεν πούμε τι είναι ειδικά η ενεργειακή αποδοτικότητα, τότε απλώς γενικόλογα θα μιλάμε για αυτήν και δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε σχέση με τη σωστή κατεύθυνση και παραμέτρους πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και δύο λόγια προς την Κωνσταντσε Κρέλ για το, τις κλιματολογικές αλλαγές και την εμπορία ρήπων ETS. Ε, ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα με τα πιστοποιητικά εμπορία ρήπων, όμως ε, πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της μείωσης εκπομπών ρήπων λοιπόν, κατά 20% και δεν έχουμε την προθυμία των κρατών μελών τα κονδύλια αυτά να τα δεσμεύσουν στη στην στοχοθετημένα στη χρήση τους αυτά τα κονδύλια τα οποία συλλέγουν από τις, τα πιστοποιητικά εκπομπών ρήπων ώστε να επενδύουν στοχοθετημένα και αποτελεσματικά. Η Γερμανία το κάνει αυτό, αλλά δεν είναι δεσμευτικό, είναι επιλογή της Γερμανίας. Αν δεν ασκήσουμε πίεση τα κράτη-μέλη να δεσμεύσουν τα κονδύλια αυτά στη χρήση τους στην, ε, ε, στοχοθετημένα μόνο για αυτή τη χρήση τότε δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει. Να δημιουργηθεί μια νέα πηγή κονδυλίων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη δεν είναι το νόημα έναντι της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό και διακυβεύει την ανταγωνιστικότητα της συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι πολύ σημαντική. Και δίνει και ένα ισχυρό επιχείρημα ε, ως προς το γιατί τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να υποστηρίξουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θεωρούσαμε μαζί με την Κομισιόν ότι οτιδήποτε κάνουμε στα πλαίσια της ε, έκθεσής μας να είναι υποφελές για την κλιματική αλλαγή. Οι μόνες των κτηρίων είναι ένα τμήμα της λύσης. Δεν είναι η πλήρης λύση. Πρέπει να μονώσουμε και τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια, αλλά θα πρέπει επίσης να προσέξουμε και τι κάνουν οι... τι γίνεται με την θέρμανση, με την ψήξη, με τα δίκτυα διανομής της ενέργειας, ο, με όλους αυτούς τους συντελεστές. Όλα αυτά τα στοιχεία εντάσσονται στα Ταμεία Συνοχής και στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν ίδιε διατάξει. Αυτό είναι καλό γιατί οι κανόνε έτσι είναι πιο απλοί για τους ε, δικαιούχου. Δεύτερον, τονίσαμε ιδιαίτερα την ε, αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα. Όχι οποιαδήποτε μορφή παραγωγής ενέργειας, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή, ε, ένας νέος τρόπος παραγωγής ενέργειας που μας εξασφαλίζει εξοικονόμηση. Αυτό είναι μια νέα φιλοσοφία, μια νέα προσέγγιση για μια νέα γενιά ε, ενέργειας, θέρμανσης και ψήξης για τις κοινότητές μας, τις κοινωνίες μας. Και τέλος, πολύ σημαντικό, όταν επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μην ξεχνάμε ότι και αυτό είναι τμήμα του συνολικού πακέτου, της συνολικής προσέγγισης. Το θέμα είναι πώς θα τα καταφέρουμε καλύτερα στο μέλλον. Θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα, θα πρέπει να δούμε πώς θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα, ούτω ώστε στο τέλος όλη αυτής της προσπάθειας όχι να έχουμε μόνο εξοικονόμηση, να έχουμε βελτίωση, αλλά να τη μετράμε κιόλα. Και κάθε κτίριο το οποίο υποφελείται από τα ταμεία του από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής και Περιφερειακής Ανάπτυξης να έχει ένα πιστοποιητικό το οποίο θα λέει ε, ποιος είναι ο ενεργειακός συντελεστής του. Έτσι είναι πολύ σημαντικό για να ετοιμάσουμε το δρόμο για μια νέα γενιά κτηρίων. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Διάφορα πράγματα ακούσαμε που μας τραβάνε την προσοχή. Καταρχάς ακούσαμε ενδιαφέροντα νούμερα για την απορρόφηση. Γιατί έχουμε αυτά τα νούμερα, είναι το ερώτημα. Άκουσα την παρουσίαση των καλεσμένων μας, ενδιαφέρουσα. Αυτό που δεν μας είπαν είναι γιατί διαφέρουν τα ποσοστά απορρόφησης τόσο πολύ. Εγώ, όπως είπε και ο Ρίχαρντ, Πιστεύω ότι αυτή η ευρωπαϊκή δραστηριότητα είναι καλή για την οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο για να την εφαρμόσουμε. <clears throat> Αυτό που δεν ακούσαμε όμως από τους ομιλητές μας είναι πόσο επηρεάζει η νομοθεσία για τις ε, κρατικές προμήθειες και πόσο υπεύθυνη είναι για τη χαμηλή ως ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης δεν ακούστηκε τίποτα για την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα, Φερρυπίν. Μέσω Φερρυπίν εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας και ελπίζω στις επόμενες παρουσιάσεις να ακούσουμε και άλλες λεπτομέρειες. Κομισιόν, όταν ακούσουμε το σχέδιο έκθεσης και είναι και εδώ ο εισηγητής, τότε θα ακούσουμε την Επιτροπή. Αρνούμε λοιπόν ομά να της δώσω το λόγο. Επομένως, θα δώσω μισό λεπτό ανά άτομο στους ε, προσκεκλημένους μας, αν μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, μην επαναλάβετε τα όσα είπατε. Υπάρχουν πολλά που έχετε ήδη πει. 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ για αυτά. Γι' αυτό που είπε η κυρία Κλέβα για το Ευρωπαϊκό ε, Ελεκτικό Συνέδριο. Ε, αυτή η έκθεση αφορούσε τα δημόσια κτίρια, που είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία από τις ιδιωτικές ε, κατοικίες, για τρεις λόγους τουλάχιστον. Καταρχάς, τα νίκια, μπορεί να χρησιμοποιήσεις τα νίκια για να εξοικονομήσεις, για να πληρώσεις μάλλον το κόστος, τμήμα του κόστου. Επίσης, ε, η σχέση κόστους-οφέλους. Ε, τι, τι επίπτωση έχει αυτό στις ε, θέσεις απασχόλησης λοιπά; Το ελεγκτικό συνέδριο δεν τα κοιτάζει αυτά. Επομένως, δεν καταλάβατε ποια είναι η αιστίαση αυτής της έκθεσης. Ε, η έκθεση ε, τονίζει σημαντικά πράγματα, ε, αξιολόγηση των αναγκών, εξάντε και εξπόστ και ποια είναι η επιλογή του σωστού επιχειρηματικού μοντέλου. Επίσης, ε, καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, δάνεια από τη μία και από την άλλη συμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. Ενδιαφέροντα αυτά τα εργαλεία, αλλά ισχύουν μόνο για ορισμένα κτίρια και ορισμένα είδη κατοικιών. Θα πρέπει να δούμε το μείγμα λοιπόν ανάμεσα σε, αυτό το, σε αυτά τα εργαλεία και στις επιχορηγήσεις που είναι πολύ σημαντικές επίσης ε, ειδικά για τις πιο φτωχές οικογένειες ή για τις, ε, τους χαμηλούς εισοδηματίες. Για την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου ακόμα ένα σχόλιο. Η έκθεση ξεκαθαρίζει ότι πολλά στοιχεία από τις, έγιναν μάλλον ανακοινήσεις για τη βελτίωση συνολικά των κτίριων και μερικές φορές δεν χρειαζόταν να γίνουν ε, επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. Θα πρέπει να έχουμε δείκτες ε, οι, οποία, οι οποίοι εστιάζουν στα αποτελέσματα, στα αποτελέσματα, έτσι, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στα νούμερα. Επίσης, τα οικονομικά εργαλεία είναι ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι είναι οι διάφοροι δικαιούχοι, θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορα μέτρα, θα πρέπει ε, να συνδυάσουμε δάνεια και επιχορηγήσεις. Ε, μιλάμε για τεχνική αρρωγή. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολύ σημαντικό, ε, είναι προτεραιότητα στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στην Τσεχία έχουμε ένα ταμείο ειδικά για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειριών, το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ε, οι τιμές ε, των ETS ε, πέφτουν και η Τσεχία τροφοδοτεί το Ταμείο Πράσινης Ανάπτυξης Ε, τα κτίρια ε, κάνουν και αυτά, συνεισφέρουν και αυτά στην όλη προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Πρέπει να το δούμε αυτό στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για την, ε, το μετρήσιμο της κλιματικής αλλαγής. Ε, εμείς εισάγουμε 300 88 ε, δισεκατομμύρια προϊόντα μάλλον ε, ορυκτά καύσιμα που αξίζουν 388 δισεκατομμύρια. Τα εισάγουμε από το εξωτερικό. Αν το μειώσουμε αυτό το ποσοστό θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια. Αν δεν έχουμε ανάγκη να εισάγουμε τόσο πολύ δηλαδή. Τώρα για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Τα εθνικά σχέδια δράσης είναι η αρχή του σχεδιασμού Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό παντού. Μερικές φορές τα σχέδια δράσης λείπουν. Επίσης, μερικές χώρες ασχολούνται πάρα πολύ με την ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως η Τσεχία, ας πούμε, ε, που έχει δώσει προτεραιότητα εκεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα με χρηματοδότηση διαφόρων τομέων. Δύο-τρία σχόλια για την κατανομή των ταμείων και την απορρόφηση. Η κατανομή ήταν 3,5 ε, η απορρόφηση ήταν 3,8. Πώς θα το μετρήσουμε, λέτε αυτό, ήταν το ερώτημα. Δεν, δεν μπορούμε, γιατί στα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις χώρες μιλάνε για την απορρόφηση. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε μια ηχνηλάτηση των αποτελέσματων, να δούμε δηλαδή από που, ότι καταλήγουν εδώ, αλλά από πού ξεκινάνε. Δεν μπορούμε να δούμε όλη την πορεία. Ε, στα στοιχεία που μας δίνουν οι χώρες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πολύ σύντομα. Αναφέραμε κάποιοι ε, κάποιους δείκτες που πρέπει να δούμε και είναι αυτοί που δείχνουν τις πραγματικές εξοικονομήσεις ενέργειας, όχι το, την έκταση που έχει η μόνωση. Τα δημόσια κτίρια δεν μας απασχόλησαν εδώ, επειδή μας είχαν πει ότι θα αναφερθούμε μόνο στα, ε, στις εργατικές κατοικίες. Βεβαίως και η ενεργική αποδοτικότητα είναι πολύ σημαντική και σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αν ε, πρέπει να μιλήσουμε γενικά για την ενεργειακή απόδοση, θα μας πάρει πάνω από μια μέρα για να το εξαντλήσουμε το ζήτημα για την ε, τοπική νομοθεσία. Πράγματι είναι ένα ζήτημα, αναφερθήκαμε στο παράδειγμα της Βουλγαρίας, όμως η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να βρει τρόπους να λειτουργήσει παρά την ε, εθνική νομοθεσία σε κάποιες περιπτώσεις. Και πάλι χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αν το αφήσουμε απολύτως ε, στα κράτη-μέλη, πολλά από αυτά δεν θα επιλέξουν ε, να παλέψουν για τους ε, στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020 και πέρα από αυτό. Κάποιες χώρες θα επενδύσουν σε μεγάλης κλίμακας και εύκολα στην εφαρμογή τους προγράμματα. Και αυτό σημαίνει ότι βάζουν τσιμέντο και άσφαλτο όσο μπορούν περισσότερο και έτσι σπαταλούν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μετά, χρηματοδότηση σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Και εδώ πέρα συμφωνώ με την ιδέα ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανοιχτή για όλους τους τομείς στέγασης και ενεργειακής απόδοση στα κτίρια. Ακόμα και στις οικογενειακές κατοικίες όπου θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλη χρηματοδότηση σε ιδιωτική στέγαση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν ε, οικονομικά ε, μέσα που να φτάνουν σε, όλ, ε, σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θέλουμε αυτή την περιληπτική ανάπτυξη. Αυτά από πλευράς μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για να κλείσουμε αυτό το σημείο της μέσης διάταξης. Την επόμενη φορά θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα θα θέλαμε να περάσουμε στο τελευταίο τμήμα της Επιτροπής μας, της συνεδρίασής μας για τον Απρίλιο. Έχουμε πέντε σημεία προς συζήτηση και μία ώρα στη διάθεσή μας. Ελπίζω λοιπόν να δείξετε πειθαρχία. Ξεκινώ με την έκθεση του Λάμπερτ Βανίστερροι και της Κωνσταντς Κρέλ για ε, τον ε, Γενικό Κανονισμό. Κωνσταντς. Η Κωνσταντσε Κρέλε. Ας αρχίσω εγώ σήμερα. Έτσι είχαμε πει ότι θα ανταλλασσόμαστε, θα είχαμε εναλλάξει παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, αξιοπρόσεκτος απολογισμός εργασίας μπορεί να παρουσιαστεί. Μπορώ να σας πω ότι από την τελευταία συνεδρίαση της ομάδας μας, της Επιτροπής μας, δέκα τριμερίσια διάλογοι έγιναν και 32 συνολικά για τον γενικό κανονισμό από τότε που ξεκινήσαμε την πρώτη φορά. Ωστόσο, ήδη την προηγούμενη φορά, τελευταία φορά είχαμε πει ότι δεν προχωρούμε παρόλα αυτά όπως το επιθυμούσαμε. Και εντωμεταξύ τι βλέπουμε. Πραγματικά προσγειωθήκαμε, γίναμε πιο νυφάλιοι και ο Φανίστερ Ρόι και εγώ σε σχέση με το σύνολο της διαπραγματευτικής ομάδας. Αυτή τη στιγμή 12 κατηγορίες εκκρεμούν στη διαπραγμάτευση. Θεματολογική επικέντρωση, στόχοι, ε, περιφερική ανάπτυξη, εκπροημίου όροι και προϋποθέσεις, ε, δόσεις, τεχνική ε, συνδρομή, διαχείριση, έλεγχος, επιλεκτικότητα, επικοινωνία, μείζωνα προγράμματα, κυριότερες δραστηριότητες. Όλα αυτά είναι εν μέρη κατηγορίες που κάποτε κατά το ίμιση περίπου μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, κατά 85% είχαν εξευρεθεί συμβιβασμοί ή συμφωνούσαμε με αυτά τα οποία πρότεινε η Προεδρία και για τα υπόλοιπα όπου ναι μεν προτείνουμε συμβιβαστικές λύσεις από το Ευρωκοινοβούλιο ή ε, από, την τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δεν διαφαίνεται δυνατότητα συμφωνίας με κανένα τρόπο με το Συμβούλιο όμως. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι. Και αυτό τι είναι. Είναι ότι πραγματικά πολύ μεγάλο χρόνο δώσαμε για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και η διαπραγματευτική ομάδα, οι διαπραγματευτές πάντα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και έτσι κατέληγαν με καλή προετοιμασία στους τριμερείς διαλόγους, ώστε πραγματικά να μπορούμε να πετύχουμε συμβαστικές λύσεις. Δηλαδή, όχι μόνο οι δύο εισηγητές είχαμε συμφωνήσει και είχαμε διαπραγματευτεί και είχαμε εξετάσει τι προτείνει η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο και σχολιάζαμε όλα αυτά τα θέματα και προετοιμάζαμε συμβιβαστικές λύσεις με αυτά τα σχόλια επιστρέφαμε, τα δίναμε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Στην διαπραγματευτική ομάδα επανερχόμαστε με όλα αυτά, διότι ένα ήταν το πιο σημαντικό για όλους εμάς. Μας ενώνει η βεβαιότητα ότι εμείς επιθυμούμε η πολιτική συνοχής να τεθεί σε ένα νέο πλαίσιο και με μια νέα μορφή από την 1η Ιανουαρίου 2014 να μπορεί να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί στις περιφέρειες. Και γι' αυτό θέλουμε να ολοκληρώσουμε με κάθε τρόπο. Θέλουμε να ψηφίσουμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τον Ιούλιο, ώστε τον Οκτώβριο να περάσουμε στην Ολομέλεια προς έγκριση. Εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Τι γίνεται? Μικροφωνισμός. Ελπίζουμε με την Ιρλανδική Προεδρία να καταφέρουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Διότι και η Ιρλανδική Προεδρία μέχρι σήμερα έλεγε πάντα ότι κατά τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας η πολιτική συνοχής θέλουν να ολοκληρωθεί ως θέμα. Ωστόσο πρέπει πραγματικά να διαπιστώσουμε κάτι και να πούμε ότι τις τελευταίες εβδομάδες ουσιαστικά δεν σημειώσαμε πρόοδο. Παρότι, παρόλο που από δική μας πλευράς ε, είχαμε εξαιρετικά προετοιμάσει τους τριμερείς διαλόγους στις συναντήσεις, ιδιαίτερα χάρη στους συνεργάτες της Γραμματείας και τους βοηθούς και, τις, ε, και τους, τη γραμματεία και τους βοηθούς της ε, κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Δηλαδή μόνο η Επιτροπή και το Συμβούλιο στους τριμερείς διαλόγους ήταν καλά προετοιμασμένοι. Πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων ξεκινά η Προεδρία τότε να διαβάζει μόνο τα έγγραφα και πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα έγγραφα, έγγραφα που μέρες πριν είχαμε αποστείλει προς την Προεδρία κτλ. Διαρκώς τα ίδια προβλήματα. Είναι θέμα λοιπόν που πρέπει να συνηθίσουμε σε κάποια πράγματα και να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Θυμάμαι την τελευταία φορά το είχα πει και στην Επιτροπή μας ότι για τα σημαντικά θέματα και για τα επίμαχα θέματα όπως για παράδειγμα ποσοστά ESF ή όροι και προϋποθέσεις εκ προημίου ή μακροπροϋποθέσεις ή προχρηματοδότηση. Δεν καταφέραμε καν να προχωρήσουμε σε αυτά. Δηλαδή τι διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε αυτά που είναι πουσιώδη στοιχεία ή λεπτομέρειες ή πράγματα που σε άλλο σημείο από το Συμβούλιο έχουν ήδη γίνει δεκτά. Παράδειγμα, είχαμε το θέμα του ότι πρέπει να προσέξουμε σε συγκεκριμένα άρθρα όταν αφορούν το ίδιο θέμα με την ίδια διατύπωση γλωσσικά να τα καλύπτουμε τα προβλήματα, με την ίδια ορολογία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οριζόντιες, για παράδειγμα, παρεμβάσεις σε πέντε διαφορετικά άθρα και να χρησιμοποιώ πέντε διαφορετικές ορολογίες ή όρους δεν γίνεται. Πρέπει να είναι ένα ενιαίο πλαίσιο. Είναι δουλειά του Κοινοβουλίου να το ελέγχει και να το διασφαλίζει αυτό. Και το κάνουμε. Και το αποτέλεσμα στους τριμερείς διαλόγους το έχουμε. Ποιο είναι. Ακούει η Προεδρία τις απόψεις μας και λέει ναι, το σημειώνουμε το ακούμε, αλλά απλώ το σημειώνουμε. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά που λέτε. Πρέπει πρώτα να τα εξετάσουμε, να τα αναλύσουμε και μετά να δούμε αν τα δεχόμαστε. Είναι δυσχερέστατη η κατάσταση σε σχέση με αυτέ τι διαπραγματεύσει. Εξαντλείται ο χρόνο. Δεν έχουμε πια άλλο χρόνο. Γι' αυτό πριν δύο-τρει εβδομάδε είπαμε ήδη θέλουμε όλα αυτά σε πολιτικό επίπεδο στους τριμερείς διαλόγους να διαμορφώνονται και να ε, ε, εγκρίνονται και να προχωρούν. Ίσως οι εκπρόσωποι της Προεδρίας δεν μπορούν να το κάνουν ή δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν το γνωρίζω. Να καταλήξουν δηλαδή σε συμβιβασμούς. Και έτσι παγώνουν τα πράγματα και λιμνάζουν. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Δεν προχωράμε. Υπάρχει απόρριψη. Δεν υπάρχει χρόνος από πλευράς Υπουργού από ό,τι φαίνεται να ασχοληθεί με όλα αυτά. Και ο πρέσβης που ρητά τον είχαμε προσκαλέσει στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή σήμερα διότι μόνο το τμήμα της ε, δημόσιας συνεδρίασης ε, της, ε, κοινο, της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής είναι δημόσιο και μπορεί αυτό δημόσια να χρησιμοποιηθεί για τους πολίτες. Ψάξτε να βρείτε που είναι ο πρέσβης. Δεν είναι εδώ, δεν παρίσταται. Λυπάμαι γι' αυτό. Ελπίζω και ευελπιστώ ότι στο Λουξεμβούργο, στο Κορεπέρ αυτή την εβδομάδα, εντάξει καλό είναι αυτό να είναι εκεί, αλλά ελπίζω ότι τα μαντάτα οι ειδήσει για όσα συζητούμε σήμερα εδώ θα φτάσουν σε εκείνον παρόλα αυτά και θα τα ακούσει. Και παρόλα αυτά η πολιτική τριμερής διάλογη στο υπουργικό επίπεδο και στο επίπεδο επιτρόπου είναι σημαντικό. Και ο Επίτροπος έχει μια ολόκληρη ε, ένα ολόκληρο κατάλογο ημερομηνιών πότε μπορεί να είναι διαθέσιμο σε τριμερείς διαλόγους. Αυτή τη στιγμή δεν παρίσταται και είναι πρόβλημα αυτό αυτή τη στιγμή σήμερα και με την Προεδρία ρητά. Και το λέω ρητά με την Προεδρία. Γιατί? Διότι όπως εμείς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που επικοινωνούν και άλλοι ευρωβουλευτές ε, επικοινωνούν και συναντούμε και εκπροσώπους των κρατών μελών. Όμως ποια είναι η πείρα μας. Η εμπειρία δείχνει και οι πληροφορίες δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη ούτε καν ενημερώνονται για το πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις στους τριμερείς διαλόγους. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν καν ευκαιρία να πούν ότι δεν θέλουμε μια τέτοια δυνατότητα ε, ψήφισης, δικαιώματος ε, ψήφισης ε, και λόγω αυτής της ψήφισης ή ψηφοφορίας να αποτύχει η πολιτική συνοχής λόγω μιας άρνησης. Δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Είναι ένα γεγονός που με κάνει να διαρωτώ με να διαρωτώ με θέλει πραγματικά η Προεδρία να πετύχει η πολιτική συνοχή και να δρομολογηθεί ή όχι και θέλει να τα τροχοπεδίσει όλα. Και αν θέλει να τροχοπεδίσει και να παγώσει τα πάντα διαρωτώ με γιατί. Κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες πολλά. Κάναμε πολλά για να βρούμε συμβιβασμούς και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και στα χαρτιά και στις προτάσεις. Ένα τρίτο αυτών που έχω εγώ εδώ μπροστά μου στους φακέλους μου αυτών που διαπραγματευτήκαμε δεν προχώρησαν. Πολλοί συμβιβασμοί που είχαν υποβληθεί επειδή και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναζήτησαν μια κοινή πορεία για την πολιτική συνοχή με συμβιβασμούς και στο μεγαλύτερο βαθμό τώρα εξαρτώνται από το Συμβούλιο, δηλαδή πάρα πολλοί συμβιβασμοί έχουν επιτευχθεί και υπάρχουν. Όμως οι συμβιβασμοί αυτοί, οι συμβαστικές λύσεις είναι της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και ποτέ, καμιά φορά από την Προεδρία, ποτέ δεν επετέχθη τέτοιο συμβιβασμός από την Προεδρία ή με την Προεδρία. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε όταν την πρώτη φορά σας ανέφερα εγώ ή σας αναφέραμε εμείς για τον πρώτο τριμερή διάλογο υπό την Κυπριακή Προεδρία. Παραπονούμαστε και λέγαμε ότι μπορούν να πάνε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αλλά κάτι διαπραγματευτήκαμε τότε. Διαπραγματευτήκαμε όλο το πακέτο της δέσμης μέτρων με την Κυπριακή Προεδρία και το ολοκληρώσαμε στη διαπραγμάτευση και υπήρξε συμφωνία και ούτε καν είχαμε καταλήξει στην ιδέα να έχουμε πολιτικούς τριμερείς διαλόγους, διότι τα πράγματα προχωρούσαν. Μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε και είχαμε και χειροπιαστά αποτελέσματα. Με την Ιρλανδική Προεδρία όμως αυτή τη στιγμή βλέπω πολύ λίγες δυνατότητες να μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ότι το σαφές μήνυμα που στέλνουμε σήμερα από την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή θα το αφουγκραστούν στην Προεδρία, στην Ιρλανδική Προεδρία θα το λάβουν το μήνυμα και τις επόμενες τρεις-τέσσερις εβδομάδες θα καταλήξουμε σε επιτάχυνση των συνολικών διοργασιών και ολοκλήρωσή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Πράγματι, συμφωνώ με τις τελευταίες παρατηρήσεις της Κωνσταντς που αναφέρει ότι στις επόμενες εβδομάδες τι επόμενε εβδομάδε έχουμε τέλο πάντων. Και αν δείτε όλα τα κεφάλαια που έχουμε διατρέξει και δεν έχουν κλείσει ακόμα, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Εκεί εντάξει δεν υπάρχει και τόσο πρόβλημα. Ουσιαστικά είναι θέμα βούληση για να ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα. Και τις τελευταίες ημέρες ε, λάβαμε ενδείξεις ότι ε, όποιος και αν έρθει, υπουργό ε, ή πρέσβης, στη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου μπορούμε πραγματικά να θέσουμε επιτάπητος και να το λύσουμε. Κεφάλαιο το κεφάλαιο. Και πράγματι μέσα στον Ιούνιο θα επιστρέψουμε με αυτά τα αποτελέσματα και δεύτερον ψηφίζουμε τον Ιούλιο για τα αποτελέσματα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι ότι κρατάμε τα πράγματα ανοιχτά για πάντα υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας, αλλά και το να μην ε, κλείνουμε ποτέ το ζήτημα δεν είναι ένδειξη καλής προεδρίας. Το ξέρουν και εκείνοι. Και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουν ε, την ετοιμότητα και τη βούληση ε, να καταλήξουμε, όπως συνέβη και στην Κυπριακή Προεδρία. Πράγματι, ανοίξαμε όλα αυτά τα κεφάλαια, εκτός από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εκεί Τα έχουμε συζητήσει τόσε φορές για τις δικές μας ευθύνε, τι αρμοδιότητες. Όλα αυτά λοιπόν που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα θα πρέπει να συζητούνται μαζί μας ανοιχτά. Και αυτά τα ζητήματα δεν τα έθεσαν μπροστά μας. Για τις ε, προϋποθέσεις, το performance reserve, τις οροφές και ούτω καθεξής. Αυτό το τελευταίο λοιπόν κεφάλαιο πρέπει να ανοίξει και ευτυχώς δεν εκφράζουμε μόνο τη θέλησή μας, αλλά πολύ σοβαρά παρουσιάζονται και από την κυρία Χιούμπνερ ως ε, πρόεδρος. Και εγώ περιμένω το, ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας της αντιστροφής. Αλλιώς χάνονται οι ελπίδες μας και θα ήταν πολύ κρίμα. Αλλά γενικά εργαζόμαστε και θέλουμε να εργαστούμε στις ε, συμβάσει εταιρικής σχέση ε, για να προετοιμάσουμε και τι περιφέρειες και να έχουμε σημαντική πρόοδο. Επομένω, σίγουρα η θέληση υπάρχει από πλευρά μα. Θέλουμε να το προσπαθήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν το ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν και με την εντολή μας και να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον ε, Ιούλιο και να περάσει και στην Ολομέλεια. Γιατί ίσως επί του περιεχομένου να μπορεί να υπάρξει συμβασμός, αλλά όταν δεν υπάρχει και καμία θέληση υποχώρηση, ίσως να μην γίνει. Δεν είναι απαραίτητο σήμερα να διατρέξουμε όλα αυτά τα κεφάλαια, αλλά για την κατάσταση θα τα ακούσετε και τον Ιούνιο. και έτσι μπορούμε να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει να παρέμβει η Κομισιόν, γιατί πρόσφατα έγιναν και δύο αλλαγέ στον κανονισμό ε, και στην απόφαση ε, για το Ταμείο Ηλίας για να λάβει αυτό θέματα που ρυθμίζει το Ταμείο Συνοχής. Θα είμαι σύντομος. Ένα γενικό σχόλιο. Υποστηρίζουμε τους στόχους του Κοινοβουλίου να υπάρξει συμφωνία ε, επί Ιρλανδικής Προεδρίας και να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος το συντομότερο δυνατόν. Εμείς ο πλευράς Κομισιόν αλλά και ο Επιτροπός μου είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ε, προσπάθεια που κάνει, ειδικά στα πιο τεχνικά κομμάτια του, καονισμού, του καονιστικού πακέτου και στα οποία έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τώρα, το θέμα είναι πού κολλάει το θέμα στα πολιτικά θέματα. Εκεί πρέπει να αρχίσουν οι πραγματικέ διαπραγματεύσει. Αύριο στο Κορεπέρ τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν την μερική γενική προσέγγιση για διάφορα θέματα ε, και για θέματα που αφορούν το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζουμε από εκεί να ξεκινήσει μια επιτάχυνση στι συζητήσει. Όπως <clears throat> και όπω είπαν και οι συγητέ, αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για να υπάρξει τελική συμφωνία για το πακέτο. Για την ανεργία των νέων και τη σχετική πρωτοβουλία, να σας πω δύο λόγια. Η ανεργία των νέων φυσικά είναι ένα από τα βασικά προβλήματα, τις βασικές προκλήσεις για την επόμενη περίοδο. Ξέρουμε τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη-μέλη και η Κομισιόν ε, έκανε αυτό το πακέτο για την ανεργία των νέων, ε, το πρότεινε το Δεκέμβριο και έχει μιλήσει γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο πολλές φορές και το Συμβούλιο το Φεβρουάριο ε, του 2013 υιοθέτησε αυτή την ιδέα. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να γνωρίσει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση ε, των νέων σε ορισμένε περιφέρειες και είναι ανοιχτό σε όλες τις περιφέρειες όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων ε, ξεπερνάει το 25% και ο προπολογισμό ε, της πρωτοβουλία είναι 6 δις. Ε, εμείς ε, τροποποίησαμε στις 12 Μαρτίου τους ε, κανονισμούς ε, και θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους θα εν, μπει στην επόμενη περίοδο για τα ταμεία και όλες οι πρωτοβουλίες για τους νέους θα αφορούν νέους που δεν βρίσκονται σε φάση εκπαιδευτική, που δεν λαμβάνουν καμία κατάρτιση κτλ. Θα ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θα εστιάσω τώρα στην βιώσιμη ολοκλήρωση, ένταξη μάλλον, συγγνώμη, των ατόμων αυτών στην αγορά εργασία. Αυτό είναι ο βασικό στόχο. Η δεύτερη τροποποιητική πρόταση υιοθετήθηκε χθε από την Κομισιόν και είναι πιο τεχνική, λιγότερο πολιτική η σημασία της. Αφορά την εναρμόνιση των δομών διαχείρισης και ελέγχου του καονισμού για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, μια μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών στο Συμβούλιο είπαν ότι δεν θέλαν αυτά που πρότεινε η Κομισιόν, που είναι η ευθυγράμμιση των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης με, τα, με το σύστημα ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Η Κομισιόν είναι ανοιχτή. Ε, εμείς θέλουμε να εναρμονιστεί και να απλουστευτεί το όλο πλαίσιο, αλλά ανησυχούσαμε ότι αν το αφήσουμε αυτό για συζήτηση στο Συμβούλιο απλώς και τελικά στους τριμερείς διαλόγους, τελικά θα έχουμε τρομερές καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Ε, γι' αυτό κάναμε μια τροποποιητική πρόταση που κάνει τρία πράγματα. Καταρχάς, βάζει το EMFF στην οικογένεια της πολιτικής συνοχής. Επομένως, ε, με σκοπό τη διαχείριση και τον έλεγχο. Έτσι. Υπάρχουν ε, προσαρμογές στον κανονισμό CPR. Κάνει επίσης αλλαγές στον κανονισμό EMFF, ούτως ώστε να βγάλει ε, τα τμήματα που αφορούν τον τη διαχείριση και τον έλεγχο και που συνδέονται με την ανάπτυξη πέθρου και υπάρχουν και κάποιες τεχνικές αλλαγές αλλά και κάποιες παρεκκλήσει που έχουν εισαχθεί ούτω ώστε να κρατήσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά του EMFF. Για να διευκολυνθεί η συζήτηση, προτείναμε αυτές τις αλλαγές και ελπίζουμε το ίδιο πνεύμα να διαπνέει ε, και τα υπόλοιπα όργανα. Ευχαριστώ, Ελίζα δεν θέλω να επισέλθω στην πρωτοβουλία για τους νέους. Ήδη έχουμε διαπραγματευτεί για αυτήν στα ουσιοδέστερα. Στην Επιτροπή Απασχόλησης, ΕΜΠΛ, βρέθηκαν συμβιβασμοί. Θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γοργά ώστε να καταλήξουμε στους τριμερείς διαλόγους και να μην υπάρξει καθυστέρηση των τριμερών διαλόγων. Αυτή είναι η ιδέα που μας εμπνέει. Ναι, αλλά θα ήθελα για άλλη μια φορά να αναφερθώ στην κατάσταση των τριμερών διαλόγων στον, στην οδηγία CDR. Διότι πιστεύω ότι βλέπουμε εδώ ότι έχουμε τρελή δουλειά που γίνεται από τους, τη διαπραγματευτική ομάδα και τους εκπροσώπους και έχουμε 12 θεματολογικά πεδία που εκκρεμούν. Υπάρχουν προτάσεις αλλαγής, όλα αυτά βαίνουν εκ παραλίλου, η γραμματεία εργάζεται θα έλεγα κατά πολύ πάνω και πέρα από τα κανονικά πλαίσια εργασίας της ε, για να τα ολοκληρώσουμε. Και ολοκληρώνουμε, ξεκινά τέλεια προετοιμασμένος ένας τριμερής διάλογος και μετά τι κάνει η Προεδρία. Ξεκινά να διαβάζει τότε τα κείμενα για πρώτη φορά. Δεύτερον, τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε ότι ούτως ή άλλως ούτε καν ένα χιλιοστόμετρο ούτε χιλιοστόμετρο δεν θέλουν να αλλάξουν όσον αφορά την πρόταση συμφωνίας το οτιδήποτε και απορρίπτουν όλες τις προτάσεις του Κοινοβουλίου κάθετα και επιπλέον εμβαλωματικά να προχωρούν όπως κάνουν γραμμή ανά γραμμή, αράδα με αράδα και διαπιστώσαμε εν μέρη αυτά τα οποία προτείνει το Συμβούλιο ακόμα και απορρέουν σε μια νυχτερινή συνεδρίαση και είναι απόλυτες ανοησίες, βλακίες αυτό διαπιστώσαμε. Δηλαδή, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο. Και παρόλα αυτά το Συμβούλιο δεν υπαναχωρεί. Είναι πιο γραφειοκρατικό από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχέση με προτάσεις, τροπολογίες, συμβιβαστικές προτάσεις ή προτάσεις μείωσης της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης του γραφειοκρατικού άχθους. Είναι οι βασιλιάδες της, γεωγραφίας, της γραφειοκρατίας και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και αυτό το μήνα είχαμε τριμερούς, τριμερείς διαλόγους. Είχαμε πάντα προετοιμαστεί καλά. Είχαμε κάνει την χρήση με τον καλύτερο τρόπο, αλλά καμιά πρόοδος δεν σημειώθηκε στους τριμερείς διαλόγους. Κανονικά θα μπορούσαμε αυτούς τους τρι, τριμερείς διαλόγους να έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον κανονισμό. Δεν θα ήταν πρόβλημα και είχαμε προχωρήσει με τις τεχνικές λεπτομέρειες, είχαμε προχωρήσει, δεν θα ήταν πρόβλημα, θα εύκολα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει και θα είχαμε συμφωνήσει και θα είχαμε εστιαστεί σε πραγματικά δύσκολα θέματα από κοινού με το ERF να είχαμε μια πρόταση. Ο λόγος για τον οποίο δεν τα καταφέραμε είναι η Ιρλανδική Προεδρία που λέει όχι κύριοι δεν είμαστε πρόθυμοι ούτε χιλιοστόμετρο ούτε εκατοστό να ανταποκριθούμε έστω. Αυτό κάνουν οι Ιρλανδοί με αυτή την τροχοπέδηση, με το πάγωμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι λοιπόν ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός των κρατών μελών κέρια σημασίας για όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Σκανδαλώδες είναι αυτό έναντι των πολιτών της Ευρώπης, των φορολογούμενων. Γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο δίλημα στο οποίο καταλήγουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε απόφαση προς έγκριση στην Ολομέλεια, που πρέπει να την έχουμε, εξαντλείται ο χρόνος. Ουσιαστικά η αρχική ιδέα μας ήταν το καλοκαίρι να έχουμε μια απόφαση προς έγκριση κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Πάμε τον Σεπτέμβριο τώρα. Όλα αυτά επειδή αυτό το σχέδιο με την Προεδρία από κοινού είχαμε συζητήσει και θέλαμε να τα πετύχουμε με λεπτομέρειες και τώρα και στη συνέχεια δεν άλλαξε τίποτα από πλευρά του. Δεν είπαν Ξέρουν και ξέρουμε ότι πρέπει το Μάιο να ολοκληρώσουμε, να έχουμε ολοκληρώσει. Και ούτε καν εκατοστό δεν υποχωρούν και δεν ανταποκρίνονται. Και όταν είπαμε, μα γιατί είναι έτσι τα πράγματα, θέλαμε τον Ιούλιο να ολοκληρώσουμε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των διαδικασιών του ήδη το Μάιο μπορεί να έχει μια συμφωνία για αυτόν τον τριμερή διάλογο. Και τότε τι έγινε. Σαν να είμαστε εμείς από το Μάιο μέχρι τις αρχές ε, Ιουλίου ή τέλη Ιουνίου σαν να υπήρχε λέει κάποια διαφορά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμιά διαφορά δεν μπορεί κανείς 32 τριμερείς διαλόγους να τους ε, καλύψει και να τους ολοκληρώσει έτσι, διότι πρέπει όταν λένε όχι ή του Συμβουλίου να ξεκινάμε από μηδενικό επίπεδο. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι που να μπορούμε να εγκρίνουμε ή να προχωρήσουμε. Μπορούμε να εγκρίνουμε κάτι και να προχωρήσουμε όταν εμείς ε, ε, δεν δεχόμαστε ε, δεν επιμένουμε στις δικές μας προτάσεις εντολής και δεχόμαστε τις προτάσεις του Συμβουλίου. Αλλά αυτό δεν έχει καμιά σχέση με συναπόφαση όταν απεμπολούμε τα δικαιώματά μας και δεχόμαστε τις προτάσεις των άλλων. Είναι, δημιουργείται μια συγκεχημένη κατάσταση παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Είναι δυσνόητο, ακατανόητο γιατί το κάνουν αυτό αυτοί του Συμβουλίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πίσω από όλα αυτά, ούτε μας γνωστοποιούν κάτι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλάζουν τα άτομα στη σύνθεση. Τα νέα άτομα στη νέα σύνθεση δεν έχουν ιδέα. Ξαναξεκινούν με την ανάγνωση των κειμένων που δεν έχουν καμία ιδέα για αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και την οποία αντιμετωπίζουμε. Και σας τα γνωστοποιώ αυτά, διότι έχω εξοργιστεί έχω θυμώσει πάρα πολύ. Προετοιμαζόμαστε καλά, με πολλή βραδινή δουλειά, νυχτερινή δουλειά που κάνουν πολλοί άνθρωποι που κάθονται κάτω και δουλεύουν και έχουν απέναντί τους αδαείς, ανίδεους. Απαράδεκτο αυτό. Και υπάρχουν και στο web stream αυτά, στο διαδίκτυο καταλήγουν να ξέρουν τι γίνεται και όταν δεν παρίστανται εδώ να μπορούν να ακούν από τις δικές μας τοποθετήσεις σε τι οφείλεται για το ότι δεν προχωράμε και δεν σημειώνεται πρόοδος και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο σημείο ξεκινάμε σε σχέση με τις περιοχές να μην μπορούν να προχωρήσουν επειδή τα πράγματα κολλάνε στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίποτα το καινούριο για τον τρομερή διάλογο. Εκτός το ότι το μόνο που λείπει είναι οι μακροοικονομικές ε, που ακόμα δεν έχει αλλάξει. Ε, δεν το έχουμε αγγίξει στο Γενικό Κανονισμό χάρη στην ε, Ιρλανδική Προεδρία και δεύτερον κοινοί δείκτες. Και πάλι είναι περίεργο. Ενώ το Συμβούλιο και η Επιτροπή το δέχτηκαν, δέχτηκαν ένα είδος συμβασμού με τους κοινού δείκτες, ε, να μπουν στο παράρτημα και μετά να υιοθετηθούν μέσω κατά εξουσιοδότησης πράξης και να μην τροποποιηθεί το παράρτημα. Ενώ λοιπόν υπάρχει συμβιβασμός και οι δύο εισηγητές, ο κύριος Όλμπριχτ και εγώ, ε, ε, στηρίξαμε αυτή τη λύση, μου είπαν ότι χθε η Ιρλανδική Προεδρία στο Συμβούλιο είπε ότι όχι, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει συμβιβασμός, ενώ υπάρχει. Και θα ήθελα να πω κάτι που συνάδει μετά σου και η Κωνσταντσα Κρέλ. Βάσει των πληροφοριών που έχω λάβει, είναι τόσο προφανές ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ της Προεδρίας και των κρατομελών, ότι δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για τη συνέχιση των τριμερών διαλόγων. Και τα κράτη-μέλη δεν, δεν ενημερώνονται ποτέ για το τι έχουμε κάνει, τι μένει ακόμα να διαπραγματευτούμε, για να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να ε, σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν και να προτείνουν λύσεις. Καμία ενημέρωση. Και αν αυτό ισχύει, τότε πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα ε, στο τέλος της διαδικασίας να εφαρμόζουν τα όσα εμείς ε, θα διαπραγματευτούμε μέσα του τριμερούς διαλόγου. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ίσως αύριο στην ΕΚΟΡΕΠΕΡ τα κράτη-μέλη να ενημερωθούν για τις εξελίξεις. Ενώ πολλά έχουν γίνει σήμερα και έχουμε πολλά επιτεύγματα στις, ε, στους τριμερούς, διαλόγους. Και πάλι, αυτό επιβεβαιώνει την πολύ κακή διαχείριση, γιατί στις διαπραγματεύσεις για τον ε, κανονισμό του Ταμείου Συνεχής, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Είχαν πολύ καλές διαπραγματεύσεις. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Και πάντα θα επικροτώ την ετοιμότητα της Επιτροπής για την εξέβρεση συμβουσμού και τη θέλησή της. Όμω εδώ βλέπουμε ότι δεν ενημερώνονται τα κράτη-μέλη καν για τις εξελίξει. Στην προηγούμενη περίπτωση που ανέφερα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ε, με τη συνεργασία μας με την Επιτροπή και πάλι όμως τα κράτη-μέλη δεν ενημερώθηκαν για τις θετικές αυτές εξελίξεις. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και τελευταίο, αν αποτύχουμε, αν δεν καταφέρουμε να υιοθετήσουμε τον κανονισμό για την πολιτική συνοχή εγκαίρως, την ευθύνη θα, πρέπει να αναλάβει το Συμβούλιο και η Ολλανδική Προεδρία, όχι το Κοινοβούλιο. Πρέπει να το ανακοινώσουμε αυτό, να το επαναλάβουμε και ίσως ακόμα και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σούλτς, ενδεχομένως να πρέπει να ε, το διαμηνήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ελληνικής Προεδρίας να τους ε, προειδοποιήσει λοιπόν ότι κοντεύουμε να αποτύχουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εγκαίρως για να προετοιμάσουμε την κατάλληλη ε, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής από το 2013. Ευχαριστούμε. Ας συνεχίσουμε ε, στο Γενικό Κανονισμό. Σον Κέλλη για τον Γενικό Κανονισμό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Και δεν είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω την Ιρλανδική Προεδρία, βέβαια. Αλλά επειδή είμαι Ιρλανδός Ευρωβουλευτής, ε, ανησυχώ για το πορτρέτο που σκιαγραφείται για την Προεδρία. Γιατί ξέρω ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση έχει πάρει την Προεδρία πολύ στα σοβαρά και γενικά είναι πολύ δεσμευμένη, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε πολλούς τομείς και νομίζω ότι αυτό που μου λέτε είναι κάτι το εξαιρετικό. Δεν, σε σχέση με τα υπόλοιπα που ακούω, είναι μοναδικό. Ο Λάμπερτ την περασμένη εβδομάδα ε, μου τα είπε αυτά ε, και όλο το Σαββατοκύριακο ε, μίλησα με υψηλού αξιωματούχου και υψηλά ιστάμενους στην κυβέρνηση. Μίλησα και χθε, μάλιστα, σε εκπροσώπους τη Ιρλανδικής κυβέρνηση και αμφισβητούν κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, με διαβεβαίωσαν ότι επιθυμούν ε, διακαώς να σημειωθεί ε, ώστε να τον προ, περισσότερη πρόοδος ε, σε αυτό το θέμα. Και αν εγώ μπορώ να βοηθήσω για να μιλήσουμε, να μιλήσετε μέσω εμού στην Ιρλανδική κυβέρνηση, πέστε μου. Αλλά πέστε μου συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Εγώ δεν συμμετέχω στον τριμερή διάλογο. Πού συγκεκριμένα υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχει φρενάρισμα, τροχοπέδι, θα το πω, γιατί πραγματικά η Ιρλανδική Προεδρία με διαβεβαίωσε ότι θέλει να σημειώσει πρόοδο σε όλους τους φακέλους, σε όλα τα θέματα που απασχολούν το Κοινοβούλιο. Και μου είπε ότι θέλει να είναι και αποτελεσματική, αλλά είναι και δεσμευμένη να κάνει καλά τη δουλειά της. Ευχαριστώ, Σον. Λουίς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου ανησυχία για τον τρόπο που τα πράγματα εξελίσσονται και κυρίως επειδή υπάρχει ένα σύνολο θεμάτων πολύ σημαντικών για τις περιφέρειες που δεν έχουν ακόμα συζητηθεί. Για παράδειγμα, οι μακροοικονομικοί όροι, για παράδειγμα για χώρες όπως την Πορτογαλία που βρίσκονται υποκαθεστώς ε, ε, υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, που ισχύει με τις μακροοικονομικές αυτές προϋποθέσεις εμείς απορρίπτουμε αλλά όταν ρυθμίζεται και αρθρώνεται με το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θέλουμε να έχουμε δι, διπλές ρυθμίσεις, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό. Μπορεί να καταλήξουμε σε καταστάσεις απόλυτα άδικες Υπάρχουν περιφέρειες στην ίδια μου τη χώρα που έχουν οικονομικές επιδόσεις καλές η ε, Τρόικα στην τελευταία αξιολόγηση για την ε, Πορτογαλία καθόρισε έλλειμμα 6,4% όσον αφορά το επίπεδο που είχε υπολογιστεί. Σε περιοχές όπως η δική μου που έχει, έχουν αυτονομία πολιτική και οικονομική είναι 0,4 το αίτημα και 19% το χρέος μόνο. Πώς μπορούν να εφαρμοστούν λοιπόν σε μια τέτοια περιοχή κυρώσεις μακροοικονομικές αυτού του είδους. Αυτά είναι παραδείγματα που οι ε, πληθυσμοί πρέπει οι, οι πολίτες δεν πρέπει να πιέζονται και να υφίστανται κυρώσεις με αυτόν τον τρόπο. Σαν να μην λαμβάνονται καν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και μετά όλα αυτά στο τέλος δημιουργούν πρόβλημα. Πρέπει στα κράτη-μέλη όταν υποβάλλονται οι εταιρικέ σχέσεις, οι συμβάσεις εταιρική σχέσης μέχρι τον Ιούνιο δεν είναι δυνατόν να απορριθμίζονται τα πράγματα τα οποία έχουν προηγούμενα συμφωνηθεί. Είναι μια διαμαρτυρία που κάνω εδώ και απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο. Απευθύνω έκκληση να παίρνει στα σοβαρά το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία συναπόφασης. Ευχαριστώ. Thank you very much for bringing also substantive issue to... Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τη συζήτηση και ε, επαναλαμβάνουμε τα όσα, επαναλάβατε τα όσα υπάρχουν για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια να την ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ένα πράγμα θα ήθελα να πω εξ ονόματος ε, της ε, προσέγγισης αυτής, για το χρονοδιάγραμμα. Θα θέλαμε τα μείζωνα ζητήματα από πολιτικής πλευράς το δυνατόν γοργότερα να αντιμετωπιστούν δεν έγινε αυτό μέχρι σήμερα. Μόνο υπουσιώδη τεχνικού χαρακτήρα θέματα εξετάζαμε. Σας ευχαριστώ. Ο τελευταίος αγορητής σε σχέση με τον γενικό κανονισμό ήταν αυτός. Θα ήθελα ένα λεπτό από τον χρόνο σας ε, να χρησιμοποιήσω, να υπενθυμίσω σε όλους ότι με την Κυπριακή Προεδρία είχαμε κλείσει. Είχαμε κλείσει αυτό. Δεν ξανά ανοίγει δεν έκρεμει ήταν πραγματικά το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη δέσμη στρατηγικά να καλυφθεί και έγινε αυτό. Αύριο θα ξανανοίξει ουσιαστικά το τελευταίο ουσιώδους χαρακτήρα ε, σημείο για τις διαπραγματεύσεις με το χρηματοοικονομικό μέσο και οι τελικές διατάξεις θα πρέπει να ανοίξουν και να διαπραγματευτούμε επ' αυτών. Για όλα τα άλλα θέματα είχαμε διαπραγματεύσεις που έγιναν, ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα από όσα διαπραγματευθήκαμε με την έννοια ότι αφήσαμε στο περιθώριο, στο πλάι ε, θέματα στα οποία υπήρχε συμφωνία και αφήσαμε ανοιχτά θέματα ε, τα οποία εκκρεμούσαν και κάποια θέματα ίσονος σημασία, όπως, ε, σημασίας όπως της περιφερικής ανάπτυξης ή και άλλα τα οποία απομένουν και που είναι πιο ουσιώδη πολιτικού χαρακτήρα κάποια από αυτά αυτή είναι η κατάσταση που θα έχουμε μπροστά μας. Αύριο θα ξεκινήσουμε με το δημοσιονομικό μέσο και έτσι λοιπόν σε σχέση με την εντολή πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία σε σχέση με τα θέματα που αφορούν το EMSF. Όχι μόνο σε σχέση με την, ε, τους όρους και ε, προϋποθέσεις για τη μακροοικονομική διάσταση, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία έχουν αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου. Αλλά επίσης και το παράτημα CSF που αποτελεί ένα θέμα που εκρεμεί για τη διαπραγμάτευση και την περιφερειακή ανάπτυξη επίσης. Ελπίζω ότι μετά από τη σημερινή Κορεπέρ, συνάντηση Κορεπέρ, θα είμαστε σε θέση να έχουμε την πρώτη διαπραγματευτική συνάντηση για θέματα EMFF και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει, θα μπορέσει να κλείσει το παράτημα και σε σχέση και με την περιφερειακή ανάπτυξη τα θέματα. Να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε ο Λαμπέρτ Φανίσελ Ρόι το σχέδιο τώρα είναι παράλληλα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να έχουμε τους τακτικούς τριμερείς διαλόγους και όλες τις άλλες διεργασίες και παράλληλα να ξεκινήσουμε τα πολιτικά δυσχερή θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν επί των οποίων δεν υπήρξε συμφωνία με την σημερινή Προεδρία μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να έχουμε ημερομηνίες από πλευράς της Επιτροπής και του Προεδρείου για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και επιθυμίες όλων. Ελπίζουμε ότι κατά τι αρχές Μαΐου θα έχουμε τους πρώτους τριμερείς πολιτικούς διαλόγους. Αυτή είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε. Και να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής. Πρόγραμμα και σχέδιό μα είναι να ψηφίσουμε προς έγκριση τον Ιούλιο και ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε αυτή την ψήφιση με γενικά συμπεφωνημένες θέσεις για το γενικό κανονισμό και σε σχέση με τις συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Ευελπιστούμε ότι παρόλες ε, τις αξιολογήσεις που έγιναν και τις τοποθετήσεις εξειδικευμένα και χειροπιαστά, ότι παρόλα αυτά, παρά τα αυτά, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο μας. Θα έχουμε και το EMFF. Για το EMFF δεν ε, θα έχουμε κάποια μεγέθη τα οποία θα μπορούν να τεθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Γι' αυτό το θέμα του κανονισμού για το EMFF έχει τη δική του σημασία. Αν θέλει να προσθέσει κάτι η Επιτροπή, αν όχι μπορούμε να προχωρήσουμε στις ε, εναπομείνασες εκθέσεις. Ε, πρώτο για το IDF παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, και αυτό το θέμα είναι πολύ πιο απλό από τον γενικό κανονισμό για τα οικοδομικά προϊόντα. Πρέπει να οριστικοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις στον τριμερό διάλογο. Το Μάιο ελπίζουμε, στις 6 Μαΐου θα είναι η τελευταία συνεδρίαση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για κάποια από αυτά τα ζητήματα, βεβαίως τα υπόλοιπα θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο πολιτικού διαλόγου. Σε ό,τι αφορά αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, υπήρξε συμφωνία για τη λεγόμενη αστική διάσταση, Urban Dimension, ιδίως ε, για αυτό το 5% της εθνικής κατανομής ε, του ERDF. Υπάρχει συνένεση για την υποχρεωτική εκπροσώπηση των αρχών στις αστικές αρχές, όμως η κλίμακα ε, πρέπει να ανέρχεται στην συνολική επιχορήγηση και νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία να μην υπάρξει αστική πλατφόρμα, αλλά ένα αστικό δίκτυο, δίκτυο ανάπτυξης για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για όλους τους συμμετέχοντες ε, για τις ε, αστικές καινοτόμες και βιώσιμες δράσεις. Αυτά έχουν συμφωνηθεί λοιπόν. Και τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν το πεδίο εφαρμογή τη ε, στήριξη, το εύρο τη στήριξη και τι προτεραιότητε επενδύσεων και αυτά έχουν συμφωνηθεί. Τι μένει ανοιχτό. Το ζήτημα των αερολιμένων συμφωνήσαμε με το θετικό στοιχείο, το περιβαλλοντικό πλαίσιο για τους αερολιμένες, αυτό είναι θετικό λοιπόν. Το αρνητικό είναι κατά πόσο θα υπάρξει αποκλεισμό εξαίρεση ε, υποδομών που δεν αφορούν ε, το περιβάλλον ή την ασφάλεια. Αλλά αυτό θα λυθεί. Για τις επενδυτικές προτεραιότητες ε, είναι το στοιχείο που ανέφερε και η Πρόεδρος χθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη λεγόμενη οικολογική καινοτομία, ε, ότι υπάγεται στον θεματικό στόχο υπαριθμών 1 και το ζήτημα της, των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προτείναμε να έχουμε πρώτον τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι το θέμα με τη θέση του Συμβουλίου. Πρέπει να αποφασίσουμε στο εσωτερικό της ε, ομάδας διαπραγμάτευσης για ε, την μετάβαση προς ε, τα ευφυή e δίκτυα αερίου και ενέργειας. Αυτό το smart gas είναι ακόμα ένα ζήτημα. Κατά την ψήφιση της εντολής δεν υπήρξε ομοφωνία. Μετά, τι κάνουμε για αυτές τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και υπηρεσίες για να, για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τους αποκλεισμούς. Και τίθεται και έμφαση στο ζήτημα των ηλικιωμένων της τρίτης ηλικίας, αλλά περιμένουμε την τελική πρόταση της ε, Κομισιόν. Το πιο επίμαχο ζήτημα είναι η θεματική συγκέντρωση. Και θα θυμάστε ενδεχομένως τους, τρεις τύπους ε, περιφερειών, ε, λιγότερο ανεπτυγμένες, μεταβατικές και πιο ανεπτυγμένες και η θεματική συγκέντρωση πάει 50-50 στις μη ε, ανεπτυγμένες, 60-40 στις μεταβατικές και στις πιο ανεπτυγμένες 80-20. Μετά τις διαπραγματεύσεις, αλλάξαμε την προσέγγισή μας και συμφωνήσαμε να διαβρινθούν οι θεματικοί στόχοι από 1-3 σε 1-3-4, ε, προσθέτοντας και το ICT. Και στην εντολή μας προτείνουμε να υπάρχει ελεύθερη επιλογή, αλλά δεν ε, συμφώνησε, δεν το δέχτηκε το Συμβούλιο. Πρόσφατα συμφωνήσαμε για κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει τουλάχιστον για δύο από τους τέσσερις θεματικούς στόχους και κάτι που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα είναι το ελάχιστο επίπεδο ε, της ε, οικονομίας ε, χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Όπως θα θυμάστε, οι θέσεις μας ήταν από την αρχή 20 για τις ε, μη και μεταβατικές και 12 για τις ανεπτυγμένες. Δεν υπάρχει συμφωνία από το Συμβούλιο. Ακόμα εργαζόμαστε για την εξέβρεση συμβαστικής πρότασης. Ελπίζω, ελπίζουμε να τη βρούμε στις 6 Μαΐου. Και βεβαίως ακόμα παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για ε, το σύνολο των εξαιρέσεων ε, που αφορά κυρίως ε, τις νησιωτικές περιοχές αλλά και τις ε, πρώην ε, περιοχές ε, phasing out να μπουν στην κατηγορία των μεταβατικών. Υπάρχει μια γερμανική, μια σπανική και δύο ελληνικές περιφέρειες και θέλουμε να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Για τους δείκτες, ο Βίκτορ το ανέφερε, προτείνουμε να μην μπει στο παράρτημα, σε αντίθεση με το ESF, αλλά να μπει ως ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Το πρόβλημα όμως ε, είναι μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής για να δουν αν θα είναι εκτελεστική ή κατεξουσιοδότηση πράξη. Όμως ε, στο, Κοινοβούλιο υπάρχει συμφωνία να προωθήσουμε κατεξουσιοδότηση πράξη και αν όχι να έχουμε το παράρτημα που θα τροποποιηθεί με την σε πράξη. 6 Μαΐου λοιπόν έχουμε τον επόμενο τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις, ακόμα και στα πιο δύσκολα ζητήματα. Και ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για την τελική ψηφοφορία θα παραμείνουν κάποια σημεία προβληματισμού ε, ε, από κάποιες πολιτικές ομάδες ε, εντός της Επιτροπής μας, αλλά βεβαίως εδώ έχουμε πλειοψηφική ψηφοφορία και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ακολουθήσουμε τους στόχους μας. Να ανοίξουμε όλα τα σημεία τώρα. Η Έρικα Μάνερ θα παρουσιάσει το δικό της. Ε, Βίκτορ, αν θες να προσθέσεις κάτι. Ε, μετά ο Ιωακίμ και μετά θα συζητήσουμε όλα μαζί, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για σε σχέση με την εδαφική συνεργασία. Επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ πως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα άρθρα 3 και 4 γεωγραφικό εύρος και θέματα κονδυλίων. Την πέμπτη θα έχουμε τον επόμενο τριμερή διάλογο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και ο τελευταίος τριμερής διάλογος ελπίζουμε ότι θα διεξαχθεί κατά τις αρχές Μαΐου όπου υποθέτουμε ότι θα έχουμε την απόφαση επί όλων των άρθρων. Είναι δύσκολα τα θέματα τα δημοσιονομικά για τα κονδύλια. Το είδαμε και την τελευταία φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να δώσει μάχη μέχρι συστάτων, ώστε η εδαφική συνεργασία στα ποσοστά της να αυξηθεί κάπως όσον αφορά τις αρχικές προτάσεις από το Συμβούλιο. Πρέπει όμως να δεχτούμε εδώ ότι... Να δεχτούμε λέω, ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να βρούμε από πού θα αντληθούν τα, αυτά τα κονδύλια όταν θα υπάρξει μια τέτοια αύξηση ποσοστών ε, όπως επιθυμούμε. Αυτό είναι μια συζήτηση που θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα. Σε σχέση με τα κονδύλια για το πρόγραμμα αυτό όπως τα ζητήσαμε από το Ευρωκοινοβούλιο θα εξετάσουμε αυτή την πτυχή. Θα εξετάσουμε και για τα δύο άρθρα την κατάσταση ξεκινώντας από σήμερα και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να ρεαλιστικά να προχωρήσουμε και για τα άρθρα 5 και 6 ουσιαστικά τα καλύψαμε αυτά στα ουσιοδέστερα στοιχεία τους όσον αφορά τις προτεραιότητες για τις επενδύσεις που καθόρισε το Κοινοβούλιο και κατέθεσε πολλές τροπολογίες για να αυξηθούν τα αριθμητικά μεγέθη. Όμως έπρεπε να δούμε αυτά τα οποία καλυπτόντουσαν ήδη από το ERDF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μόνο τα πολύ εξειδικευμένα θέματα προτεραιοτήτων στην εδαφική συνεργασία είναι εκείνα τα οποία θα εντάσσονται στα πλαίσια αυτού του κανονισμού. Δηλαδή αποδυναμώθηκαν πάρα πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό καθιστά σαφέστερη την εικόνα και ίσως πιο εύκολα τα επιχειρήματα τα οποία τίθενται από πλευράς μας. Τελευταίο τώρα, θεματολογική επικέντρωση, άρθρο 5. Έχουμε μακρές συζητήσεις που διεξήχθησαν σε σχέση με αυτό το θέμα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 80% για τέσσερα θέματα και 20% ελεύθερη επιλογή όπως προτείνεται από το Συμβούλιο είναι κάτι αποδεκτό. Δηλαδή συμφωνούμε όσον αφορά το βαθμό ελαστικότητας μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Όμως έχουμε δύο τριμερείς ε, διαλόγους και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο Βίκτορ παρακαλώ. Ο επόμενος ε, τριμερής διάλογος θα γίνει 13 Μαΐου και μάλλον θα είναι ο τελευταίος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε αν στον τριμερή διάλογο το CPR θα υπάρξει πρόοδος για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Το λέω ξανά και ξανά. Μας είπε το Συμβούλιο ότι επιμένει στις μακροοικονομικές προϋποθέσεις και ένας μεγάλος αριθμός κρατών μελών αντιτίθενται στεναρά, αλλά δεν ενημερώνονται από την Προεδρία όμως. Το έχω πει 100 φορές. Ε, το δεύτερο θέμα είναι αυτό των κοινών δικτών που ανέφερε και ο κύριος Όλμπριχτ πριν. Υπάρχει μια πολύ εύκολη λύση να φτάσουμε σε ένα καλό συμβιβασμό, αλλά η Ιρλανδική Προεδρία αναβάλει την εξέβριση λύσης. Χωρίς το συμβιβασμό για τους κοινούς δείχτες, Έχουμε πρόβλημα με το Ταμείο Συνοχής, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εδαφικής Συνοχής και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γιατί αποφασίσαμε να έχουμε τους ίδιου δείκτες και στα τρία ταμεία αυτά και στους τρεις κανονισμούς των ταμείων. Είναι κοινοί οι δείκτες. Πρέπει να σεβαστούμε την εντολή μα. Να υπάρξει συνοχή και να δώσουμε δυνατότητα να υπάρξει πιο εύκολη εφαρμογή και καλύτερη παρακολούθηση από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Γι' αυτό κάνουμε ξανά έκκληση στην Ιρλανδική Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί και να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Αν υπάρξει πρόοδος μέχρι τα μέσα Μαΐου, θα είναι καλό αυτό. Τότε θα ολοκληρώσει η ομάδα μου τις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Συνοχής και το σχετικό κανονισμό. Ε, και θέλω εδώ να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου της διαπραγματευτικής ομάδας. Ο Γιώργη, με ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, και στη δική μου περίπτωση δεν υπάρχουν πολλά καινούρια υπό τον ουρανό των Βρυξελών από την τελευταία φορά. Ξεκινήσαμε με ορμή τις διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία καταλήξαμε στα παιδινά και κολλήσαμε και η εντύπωση που έχω είναι ότι για το Συμβούλιο λιγότερο η εκπροσώπηση της, του Συμβουλίου διαπραγματεύεται και περισσότερο διαπραγματεύονται οι εκπρόσωποι του νομικού, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Καταλήγουμε από το ένα δοκισίσοφο θέμα στο άλλο δοκισίσοφο θέμα των νομομαθών. Και σε σχέση με τα θέματα αυτά επιβαρύνεται η πρόοδος και η διαδικασία. Σε σχέση με τους ε, ετούντες για το πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλίζονται τα πράγματα να είναι το δυνατόν απλούστερα και πιο εύκολα για την, επιχειρήσει. τις επιχειρήσεις. Υποθέτω ότι η θέση του Συμβουλίου είναι να δυσχεράνει όλο και περισσότερο τις ε, θέσεις που προτείνει το, το Κοινοβούλιο και να επιβαρύνεται όλο και περισσότερο η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Ένα ολόκληρο σακί ετοιμάτων των κρατών μελών έχει το Συμβούλιο που δύσκολα μπορούν να συναρτηθούν το ένα με το άλλο και κολλάμε στα ίδια ζητήματα. Θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, για παράδειγμα προσλήψεων, εξακολουθούν να μην αποσαφηνίζονται και να μην υπάρχει μια βιώσιμη αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Η πρόταση του Κοινοβουλίου για παράδειγμα και αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρακτική να αντλούμε αυτό που πρέπει να γίνει και που είναι σωστό. Κράτη-μέλη όμως όπως η Γαλλία λένε ότι Γάλλοι υπάλληλοι πρέπει να ε, ενταχθούν σε αυτή την υπηρεσία και να έχουν δικαιώματα προσωπικού που θα είναι γαλλικού χαρακτήρα, γαλλικού δικαίου. Παράλογο είναι αυτό. Εκείνοι που θα προσλαμβάνονται από αυτόν τον οργανισμό να αποφασίζουν με ποια κριτήρια θα προσλαμβάνονται και τι θα ισχύει για αυτούς. Επίσης όσον αφορά το θέμα της διεύρυνσης ε, αυτού του οργανισμού όσον αφορά τρίτα κράτη. Τίθεται εδώ το θέμα ποια είναι αυτά τα τρίτα κράτη και κάνουμε λόγο εδώ για γειτονικέ χώρες, όμορε όμορες χώρες ε, σε σχέση με την ΕΕ. Και πάλι δεν είναι απόλυτα σαφές ποια είναι αυτά τα κράτη που είναι γειτονικά κράτη. Είναι εκείνα τα κράτη που έχουν μέσα γειτονίας που λειτουργούν ήδη για αυτά ή γεωγραφικά κοντινά κράτη, γειτονικά κράτη και αυτού του είδους ε, προβλήματα υπάρχουν. Μετά το θέμα της ε, αδειοδότησης με την προθεσμία έξι μηνών εξακολουθεί να είναι επίμαχο αυτό το θέμα. Οι νομικές υπηρεσίες ε, συνήθαν και συνεργάστηκαν πριν από τρεις ημέρες για παράδειγμα υπέβαλαν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που θα είναι η βάση τώρα ενός επόμενου τριμερούς διαλόγου. Εκείνο που είναι δύσκολο όμως είναι να βρεθούν σωστές ημερομηνίε για την γενική ρύθμιση, για το γενικό κανονισμό όταν είχαμε 32 τριμερούς διαλόγους που διεξήχθησαν ήδη και όταν βλέπουμε ότι είναι περιορισμένα τα στελέχη της Ιρλανδικής Προεδρίας από πλευράς δυναμικού και έχουμε και άλλα στοιχεία κανονισμών που είναι υποσυζήτηση, μπορώ να δείξω εν μέρη κατανόηση για αυτή την κατάσταση των πραγμάτων παρότι δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου ότι τώρα θα πρέπει να αναμείνουμε για μια νέα τέτοια ημερομηνία να μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Γιατί η συζήτηση για το γενικό κανονισμό και σε εμάς όλο και πάλι είχαμε εμπλοκή και επίπτωση από αυτή την κατάσταση. Σεβασμό πρώτα απ' όλα όσον αφορά τους εισηγητές και το, το προσωπικό και συνεργάτες και της γραμματείας και της νομικής μας υπηρεσίας που έκαναν τεράστια δουλειά, γιγάντια δουλειά βλέποντας τα, τα διάφορα πρότυπα τα οποία εξετάστηκαν και αναλύθηκαν. Ερώτησή μου, το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε μπροστά μας τώρα και το οποίο θέσαμε εμείς μπροστά μας εξακολουθεί να μπορεί να τηρηθεί. Μπορεί να τηρηθεί ή όχι όταν όλα είναι ανοιχτά και τίποτα δεν έχει αποφασιστεί και όλα εκκρεμούν και οι, μακροπροθε... οι προ όροι και προϋποθέσεις ε, για τη μακροπρόθεσμη ε, αντιμετώπιση. Τι θα αποφασίσουμε τον Ιούλιο όταν όλα αυτά εκκρεμούν. Θα έχουμε μια δική μας ξεχωριστή γνωμοδότηση, ένα σχέδιο κανονισμού που δεν θα έχουμε συμφωνήσει επ' αυτού με το Συμβούλιο και τι θα γίνει μετά στη συνέχεια. Πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα δεδομένης της κατάστασης και σε σχέση με το άνοιγμα του αεροδρομίου του Βερολίνου είχαμε αρνητική ε, εμπειρία είδαμε πολλά αρνητικά πράγματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ξέρω ότι η πίεση από τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα λειτουργικά τους προγράμματα τα κράτη και οι περιφέρειες πρέπει να υπάρξει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Αυτά όμως ε, τα οποία προτείνει το Συμβούλιο δεν μπορούμε χωρίς αντιρρήσεις να τα δεχτούμε και ενώ έχουμε δουλέψει πάρα πολύ να απεμπολίσουμε δικαιώματα και θέσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέσσερις έχουν ζητήσει τον λόγο. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Πλησιάζουμε το τέρμα της συνεδρίασής μας. Παρακαλώ συντομία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά δεν θέλω όλα να τα επαναλάβω, σίγουρα όχι. Δεν θέλω να διαφωνήσω με τον κύριο Όλμπριχτ, καθόλου δεν το επιθυμώ, αλλά δεν βλέπω πραγματικά να, να αναφύεται το τέρμα των διαπραγματεύσεων, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Επί της ουσίας πρέπει να προετοιμαστούμε και να συζητήσουμε σε σχέση με την Επιτροπή μας και όταν βλέπουμε ότι πριν από μια επόμενη συνεδρίαση ε, απομένουν θέματα δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί σε σχέση με την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών και με την Ιρλανδική Προεδρία. Σωστό είναι ότι κάποια πράγματα αποφεύθηκαν όμως ε, αυτό δείχνει ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα συζητήσαμε για πράγματα επί των οποίων δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε και ένα σχέδιο δικτύωσης, ε, καλύτερο από την αρχική απόρριψη Θυμάμαι ακόμα και με τους συμβιβασμούς τι έγινε σε σχέση με τη θεματολογική επικέντρωση. Ήταν κάτι σημαντικό για μας στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να πούμε το 4 συν 1 ή 3 συν 1 να είναι ελεύθερα επιλέξιμα στοιχεία. Είπαμε εντάξει θα έχουμε 4 και ένα από αυτά θα είναι αυτό το στοιχείο το οποίο μας προτείνατε διότι στα περισσότερα κράτη-μέλη πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει η πρόταση αυτή. Συμβιβασμοί, η πρόθεση για συμβιβασμούς που ήταν δεδομένη και ανταποκριθήκαμε στο Συμβούλιο σε σχέση με ε, προτάσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν και πρέπει να ρυθμιστούν χωρίς αμφιβολία όσον αφορά τη θεματολογική επικέντρωση. Όλα αυτά όμως πριν από τον επόμενο τριμερή διάλογο θα μπορέσουμε να τα κάνουμε να τα διασφαλίσουμε. Είναι σημαντικό σήμερα αυτό το οποίο απέρευσε από τη συζήτηση σε σχέση με τις ποσοστώσεις για τους στόχους πρέπει να καθοριστούν αυτά και πρέπει να τα συζητήσουμε σε βάθος. Όπως είπα τη Δευτέρα πριν από τον επόμενο τριμερή διάλογο θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και εγώ θα το έβρισκα καλό αν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε. Όμως δεν φαίνεται να προδιαγράφεται ο τερματισμός αυτού του εγχειρήματο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες το προσωπικό και από την ομάδα που είναι καλή ομάδα ακόμα και αν το ένα ή το άλλο σημείο έχει δημιουργεί κάποια προβλήματα. Ευχαριστώ. Μαντέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ελπίζω να καταφέρουμε να υπάρξει τελική συμφωνία ήδη στις 6 Μαΐου στον τριμερή διάλογο. Αλλά το να κλείσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ότι θυσιάζουμε τα ουσιαστικά σημεία της εντολής μας. Και ένα από τα ουσιαστικά σημεία της εντολής μας είναι η θεματική συγκέντρωση και πιο συγκεκριμένα ε, ο στόχος 4, ε, που είναι μια οικονομία ε, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Εκεί υπάρχουν προγράμματα βιώσιμων μεταφορών που απορροφούν σημαντικά ποσά. Η Κομισιόν μας υποστηρίζει στην ιδέα ότι πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά για κάθε μία από τις ε, κατηγορίες των περιφερειών δεδομένου της σημασίας της ε, οικολογικής πρόκλησης και στις ε, ανεπτυγμένες περιοχές αλλά και στα νέα κρατημέλη. Όπως έδειξε και η συζήτηση που κάναμε. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον το 22% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενεργειακή αποδοτικότητα στις αντιγμές περιοχές και στις μεταβατικές περιοχές. Ε, το 12% ε, του ποσοστού, το 12% του ταμείου για τις λιγότερο αντιγμές περιοχές. Αυτή είναι η εντολή μας. Νομίζω ότι το Συμβούλιο μπορεί να κάνει α, κάποιες υποχωρήσεις, ε, γιατί μας υποστηρίζει και η Κομισιόν. Και αυτό είναι σημαντικό για μας. Ε, κάτι άλλο που είναι κόκκινη γραμμή για τους οικολόγους είναι το να μην ε, βάλουμε στο τελικό κείμενο τις υποδομές ε, φυσικού αερίου. Αυτό που απορρίφθηκε κατά διάρκεια της ψηφορίας μέσω της τροπολογίας, μέσω μιας τροπολογίας, δεν πρέπει να ξαναμπεί από το παραθυράκι τροποποιώντας την εντολή. Δεν γίνεται αυτό, δεν πρέπει να γίνει. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή, κυρίως για τους οικολόγους. Ευχαριστώ. Κορνέλια Χένστ. Ευχαριστώ. Τρία σημεία. Πρώτο, πραγματικά πρέπει κάποια πράγματα να τα συμφωνήσουμε, να τα εντάξουμε στον γενικό κανονισμό σε σχέση με την αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Κατά πόσον αυτά μπορούν να ενταχθούν σε ένα γενικό κανονισμό δεν είμαστε βέβαιοι. Υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστούν κάποια πράγματα. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Το πρώτο είναι η θεματολογική επικέντρωση κατά κάποιο τρόπο από τον ήπιο τείχο, το, την ήπια αντιμετώπιση, καταλήγουμε στη σκληρή αντιμετώπιση με το Συμβούλιο όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα αυτά τα οποία μας προτάθηκαν δεν είναι δυνατόν να μας ε, οδηγήσουν στο να προχωρήσουμε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θέλουμε τους δικούς μας στόχους που εμείς ε, τους αποφασίσαμε και εγκρίναμε πολλαπλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπάρχουν οδικές οδικοί χάρτες, υπάρχουν προγράμματα δράσης. Όλα αυτά θα τα αγνοήσουμε, θα τα παρακάμψουμε ή θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτά. Πρέπει να δώσουμε μάχη, θα έλεγα, η ενεργειακή αποδοτικότητα να μην εξαλειφθεί, να μην απαλληφθεί, να μην καταλήξουμε σε ένα παζάρι ανατολίτικο εδώ, για ένα παζάρι με το Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο δεν έχουμε εντάξει στις ε, ε, προτεραιότητες για τις επενδύσεις από πλευράς εντολής ε, την FEE, αυτή προσέγγιση και πρέπει να μην συγχαίουμε τα πράγματα σε σχέση με την εντολή. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να υποστηρίξουμε τις υποδομές ή τις δομές. Δεν χρειάζονται πάντα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά. Δεν παρακολύουμε στα κράτη-μέλη να προαθούν αυτές οι υποδομές. Αυτό μπορούν να τα κάνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Όμως ε, κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δεν πρέπει να συγχέονται εδώ. εδώ έχουμε κόκκινες γραμμές από αρκετές κοινοβουλευτικές ομάδες που δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού ξεπερνώντας αυτές τις ε, κόκκινες γραμμές να σπάσουμε τη συμφωνία επί της οποίας είχαμε τοποθετηθεί θετικά αρχικά. Ευχαριστώ. Η Ρίκα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θέλω να μιλήσω για κάποιες ε, προτεραιότητες του, των φιλελεύθερων. Καταρχάς, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτέ αυτές ενδιαφέρουν πάρα πολύ την πολιτική μας ομάδα και θέλουμε να ληφθούν υπόψη. Οπωσδήποτε. Το φυσικό αέριο, επίσης, πολύ σημαντικό θέμα για μας. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα τα χρήματα αυτά να ε, χρησιμοποιούνται για το έξυπνο φυσικό αέριο, για τη θεματική συγκέντρωση και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, 22% για τις ανεπτυγμένες περιοχές και τις μεταβατικές περιοχές. Αυτό είναι ένας ε, υγιής και φιλόδοξος στόχος και 12% για τις χώρες συνοχής. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή του συνεργασία. Αυτά ήθελα να πω για τις προτεραιότητε των φιλελεύθερων. Για τις χώρες που έχουν ενεργειακές υποδομές τεράστιες όπως η Πολωνία, ε, το 95% του ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται από άνθρακα. Επομένως, ε, ο στόχος της ε, οικονομίας χαμηλών εκπομπών είναι δύσκολος. Λουίς, έχει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και μια και φτάσαμε στο τέλος να απευθύνω μια έκκληση στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας στην Ευρώπη προς τη συνάδελφο Ρίκε που έχει επιληφθεί του τριμερούς διαλόγου για το άρθρο 3 που κάνει λόγο για τη γεωγραφική κάλυψη. Εδώ, σε σχέση με τις ε, περιφέρειες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της... Ε, από την απόσταση 150 χιλιόμετρων ε, θαλάσσια απόσταση. Όλα αυτά όμως ε, θα πρέπει να τα δούμε στο σωστό πλαίσιο. Θέλουμε νησιωτικές περιοχές που έχουν μεγάλη απόσταση από τα ε, χερσαία σύνορα που είναι τα μεγαλύτερα, μεγαλύτερη απόσταση από 150 χιλιόμετρα θα έπρεπε και αυτές να ενταχθούν σε σχέση με αυτόν τον αποκλεισμό. Ίσως θα μπορούσαν να εξεταστούν πώς θα αντιμετωπιστούν για την, Μαδέρα ή τις Αζόρες που έχουν τέσσερις φορές σε σχέση με το πληθυσμιακό κριτήριο αλλά απέχουν πάνω από 150 χιλιόμετρα και έχουν δυναμικό εδαφικής συνεργασίας πάρα πολύ μεγάλο ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάμε να ανοίξουμε μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιρίας οικονομικά από πλευρά τουρισμού όσον αφορά την έρευνα την επιστήμη, τις τεχνολογίες. Άλλες νησιωτικές περιοχές όπως αυτές θα πρέπει υποδειγματικά να αντιμετωπιστούν. Και το γεγονός ότι αυτό το άρθρο που αφορά τη γεωγραφική κάλυψη θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές τις περιοχές, να τις εντάξει. Θα ήταν ένα παράθυρο που θα άνοιγε ευκαιρία για αυτές τις περιοχές. Θα ήταν καλό αυτό και για αυτές τις περιοχές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε στο τέλος της ημέρας της διάταξης. Επομένω, από πλευρά μου, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι η ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση 29 και 30 Μαΐου. Μια μισή μέρα έχουμε στη διάθεσή μας και ελπίζω να έχουμε καλές ευχάριστες ειδήσει για τις διαπραγματεύσεις. Ε, τέλος συνεδρίασης.